Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να αρχίσουμε την τελευταία μας συνεδρίαση, την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας, πριν ε, από τις διακοπές. Για όσους θα πάνε διακοπές το λέω. Εύχομαι λοιπόν καλές διακοπές σε όσους πάνε. Μόλις ησυχάσετε, λέω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Όπως είπαμε και στην έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε στο Στρασβούργο, η εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών και η έγκριση ε, του σχεδίου έκθεσης ε, του κυρίου Μπέκερ ε, για την πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αναβληθεί, έχει αναβληθεί στις, για τις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μας συνεδρίαση, για να είναι κάπως πιο περιεκτική η εξέταση νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση αυτή. Αλλάξαμε κάπως την ημερήσια διάταξη γιατί έτσι απελευθερώθηκε λίγος χρόνος και οι, δια... ήταν οι εξή. Όσον αφορά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το σημείο 18 δηλαδή, θα το συζητήσουμε σήμερα το πρωί είτε πριν είτε μετά από την ψηφοφορία, αναλόγως με το πώς θα τα πάμε από χρονικής απόψεως ε, και η έκθεση του ε, κυρίου Τόμας Χέντελ ε, για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης μπορεί να συζητηθεί μετά την ψηφοφορία και το σημείο 11, Μάκιντάιρ, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα, συζητηθούν, θα συζητηθεί πριν από το σημείο 8, δηλαδή πριν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως επίσης και η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Καλύτερα όμως πρώτα η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα και μετά η έκθεση, γιατί ούτως ή άλλως έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα ε, που θα συζητήσουμε στο πλαίσιο της προφορικής ερώτησης. Όσον αφορά τώρα το σημείο 21 της κυρίας Γκένς, σήμερα το απόγευμα θα το συζητήσουμε μετά το 17. Επειδή λοιπόν αναστατώθηκε η μερίσια διάταξή μας, ε, η γραμματεία θα ε, σας έχει διανύμει μία αναθεωρημένη έκδοση της μερίσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω καταρχάς ότι σε σχέση με την έκθεση της κυρίας Μπάστος ε, Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος του κυρίου Μπερλιγκέρ στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και επειδή αναβλήθηκε η έκθεση πρωτοβουλίας του και εμείς ε, αναβάλαμε και προσαρμόσαμε το χρονοδιάγραμμά μας ε, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους σας και σε όλες σας να επεξεργαστούν ε, την απάντησή τους και την επιχειρηματολογία τους, οπότε οι τροπολογίες έχουν προθεσμία πλέον μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. 19 Νοεμβρίου θα συζητήσουμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι καθυστερούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα αυτό για να μπορέσουμε στις 6 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε την έκθεση τη κυρία Μπάστο στην Επιτροπή μα, διότι η Επιτροπή Περιφερειών, Περιφερικής Ανάπτυξης ε, ψηφίζει μία εβδομάδα μετά. Θα ήθελα να σας πω και ορισμένα πράγματα. Ε, να σας καλωσορίσουμε την ε, Καμέλια Οαΐντα, η οποία δεν είναι εδώ. Ε, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι εδώ. Και στην Ιζαμπέλ Ριάννη, την βοηθό της, ε, η οποία είναι μέλος της γραμματείας από 1η Ιουλίου. Αντικαθιστά επισήμως η κυρία Οΐντα, το συνάδελφο Ματίκ να χαιρετήσουμε την Κριστίνα Βίλινσομ η οποία φεύγει από τη γραμματεία της Επιτροπής μας από 1η Σεπτεμβρίου. Α, είναι εδώ. Ξέρετε πολύ καλά τι χάνετε. Ε, από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα φύγετε, οπότε το καλοκαίρι θα συνειδητοποιήσετε τι χάνετε φεύγοντα από τη γραμματεία τη επιτροπή μα. Σα ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για όλα όσα συνεισφέρατε στην Επιτροπή μα. Επίση, βγαίνουμε και στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια δεν νομίζω να είναι κάτι το καινούριο για κανέναν. Πάμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη. Να δώσω στην εισηγήτριά μα, την Ντανούτα Γιασλοβιέσκα, την, ε, το λόγο για το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως απάντηση στην κρίση. Κυρία Συγήτρια, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Θα κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Να σας ενημερώσω λίγο για τις ε, τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε ήδη εκπονήσει και αυτό θα φανεί, ε, το κλίμα συνέντευξη δηλαδή, ενώ που υπάρχει με τους υποβάλλους τροπολογίες, άμεσα. Ε, αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφε, θα ήθελα να σας πω ότι για όλους όσου δεν συμμετείχαν στι συμβιβαστικέ τροπολογίε, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασή μα. μας Όσοι δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσει, καλό θα ήταν να γνωρίζουν ποια είναι τα κύρια σημεία των συμβιβαστικών τροπολογιών. μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε ποια είναι τα σημεία που συζητήθηκαν περισσότερα, αυτά που σα απασχόλησαν περισσότερο, για να διαφωτίσετε κάπω τη δημόσια συζήτηση. Γιατί αν μένουμε απλώς στον τύπο ή αν κάποιο παίρνει το λόγο για να πει μόνο για να πει τι καταπληκτική που ήταν οι σκιώδεις συζητητές και τι φανταστικό που είναι ο συμβιβασμό ε, και ότι θα γίνει πολύ καλή ψηφοφορία. Ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει νόημα να συνεδριάζουμε. Μην το πάρετε στραβά αυτό που σας λέω. Απλώς... έχει νόημα νομίζω η Επιτροπή, των, η Επιτροπή μας να συνεδριάζει με κάποιο περιεχόμενο. Μπορώ λοιπόν να σας ξαναδώσω το λόγο για να μας διαβοτήσετε σε 2, 3, 4, 5, εντάξει όχι 25, αλλά τέλος πάντων στα σημαντικότερα σημεία των συμβαστικών τροπολογιών για να μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση και οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Σε ό,τι αφορά τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, που ουσιαστικά αποτελούν το 8% περίπου των ε, συνολικών τροπολογιών, προσπαθήσαμε σε αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες των συναδέλφων. Η τροπολογίες αυτές πραγματικά εμπλουτίζουν το αρχικό μου κείμενο. Δεν έχει νόημα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες και να παρουσιάζω αυτές τις τροπολογίες. Απλά θέλω να πω ότι έχουμε αρκετά καλέ συμβαστικέ τροπολογίε για ένα μεγάλο μέρο αυτών και να πω ότι είχαμε και κάποιε δυσκολίε σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, η ομάδα των σοσιαλιστών ε, ήθελε πίεζε μάλλον για μια πρόταση. για μια δήλωση συγκεκριμένα στο κείμενο που εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη. Τι εννοώ. Αυτό που επιθυμεί ο Μαδός είναι τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν επαρκείς μισθούς για όλους τους εργαζομένους, επαρκής κατάλληλους μισθούς για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Εμείς διαφωνούμε με αυτή τη διατύπωση. Συμφωνούμε με το δικαίωμα του εργαζομένου να έχει ένα καλό βιωτικό ε, επίπεδο, αλλά υπάρχει και μία πραγματικότητα που αφορά κράτη-μέλη που δεν έχουν καν θεσπισμένο κατώτατο μισθό. Και να αναφερθώ και σε μία άλλη συμβαστική τροπολογία. Αποφασίσαμε να διαγράψουμε μία φράση στο κείμενο που αφορά τις συντάξεις, καθώς καλό να περιμένουμε την λευκή βίβλο για τις συντάξεις. Αυτά ήταν τα πλέον ακαθόδη ζητήματα στην ε, διεκπαιρέωση τροπολογιών και πιστεύω ότι μαζί με τους Κιώδης καταφέραμε να φτάσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Παπαδοπούλου. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, όπως και τους Κιώδης, για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έκθεση συντάχθηκε από μέλος του ΕΛΚ, θεωρούμε ότι είχε ένα πολύ θετικό τελικό αποτέλεσμα, μια τελική εικόνα, γιατί για πρώτη φορά το ΕΛΚ δηλώνει ότι τα μέτρα λιτότητας δεν αρκούν για να ξεπεράσουμε την κρίση και η εξαγίανση των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να συνοδευτεί από μια πολιτική ανάπτυξη. Μας ικανοποιεί αυτή η δήλωση. Από τις 154 συνολικά τροπολογίες, 22 συμβαστικές, θεωρούμε ότι ήταν πολύ καλή η συμπερίληψη και η αποδοχή 8 δικών μας τροπολογιών και να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα. Στην συμβαστική τροπολογία D ε, επικρίνουμε τα προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας, καθώς η οι στόχοι μάλλον κοινωνικής, πολιτικής και παιδείας ε, στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 δεν έχουν ε, αντιμετωπιστεί επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ότι αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Έπειτα, στην συστηματική τροπολογία X, καλούν τα κράτη-μέλη να προσεπογράψουν ένα κοινωνικό σύμφωνο που να περιέχει ένα ελεκτικό μηχανισμό ώστε να ανταποκριθούμε στους στόχους κοινωνικής πολιτικής και παιδείας της στρατηγικής 2020. Ε, Στην συμβασική τροπολογία Β ε, είχα μακρά συζήτηση. Θέλαμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο ορισμό ε, του όρου ε, κοινωνική διακυβέρνηση. Η κοινωνική διακυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έναν πολύ δυναμικό και ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης των κοινωνικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων του 2020. Στην συμβασική τροπολογία Β αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση της, κοινωνική, της οικονομικής συγγνώμη, εξάρτησης και ζητούμε να μην υπάρξει άμεση σύνδεση της αύξησης ε, του προσδόκιμου ζωής ε, με τα όρια ταξιοδότηση όπως ε, αρχικά απαιτούσε το ΕΛΚ. Στην τροπολογία M καλούμε για αηφόρες θέσεις εργασίας για άνδρες και γυναίκες. Τέλος, άλλες δύο ακόμη τροπολογίες θέλουμε να αναφερθούμε στην U. Μιλάμε για μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία στην αγορά εργασίας και στην R ζητούμε καλύτερα στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές σε αντίθεση με τα μέτρα α, εργασιακής ενεργοποίησης, όπως αρχικά ανέφερα στο κείμενο. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι με αυτές τις τροπολογίες καλύπτει η θέση μας, γι' αυτό προτείνουμε την υπερψήφιση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω επίσης και όλους τους κοιόδης και ιδίω την εισηγήτρια για τη βοήθεια που μου παρήχαν ε, προσωπικά και ιδίω ο κύριος Γιάνκος, ο γραμματέας του SND. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Όχι. Μπορούμε τότε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. πιο μετά θα ψηφίσουμε. Πάμε τότε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Να δώσω το λόγο στην Εμέρ Κοστέλιο για την εξέταση των τροπολογιών της ε, έκθεσής της ε, για ε, την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής για το 2011. Κυρία Σιγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρουσιάσαμε το σχέδιο γνωμοδότησης στην πρώτη συνεδρίασή μας στις Βρυξέλλες. Έγινε αρκετά βραχυπρόθεσμα και κατάλαβα ότι οι συνάδελφοι είχαν ελάχιστο χρόνο για να υποβάλουν τροπολογίες. Πάντως εννέα κατατέθηκαν και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες και τις προτάσεις τους αυτές που εν πολλής βελτιώνουν το σχέδιο γνωμοδότησης και με χαρά τις δέχτηκα τις τροπολογίες αυτές που υπογραμμίζουν τις κοινωνικές πτυχές θετικής συνοχής ασχολούνται με την ισότητα των φύλων, την εργασία των μεταναστών εντείνουν, δυναμώνουν τις κοινωνικές ρήτρες που θέλαμε να τις αναδείξουμε ιδιαίτερα για να δείξουμε την κοινωνική αλληλεγγύη στην αγορά εργασίας, αλληλεγγύη, ε, αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Λοιπόν, ε, νομίζω γενικά ότι όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν βελτιώνουν την αρχική γνωμοδότηση και με χαρά θα τις δεχτώ. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό βήμα και είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να παρουσιάσει μια αρκετά στιβαρή γνωμοδότηση για την πολιτική συνοχής. Εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους ειδικού και γενικούς στόχους της συνθήκης του Μάστριχτ από το 1992. Οπότε τις καλωσορίζω. Τώρα για τον κατάλογο ψηφοφοριών, από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μια πρόταση να αφαιρεθεί η λέξη binding, δεσμευτική, από τη γνωμοδότηση. Και νομίζω ότι η ιδέα της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, όταν αποφάσισε να γνωμοδοτήσει, ήταν να είναι στιβαρή, στεναρή γνωμοδότηση με υποχρεωτικές διατάξεις, δεσμευτικές και απογοητεύομαι που υπάρχει αυτό, αυτή η κίνηση να βγει λέξη binding δεσμευτική από τη γνωμοδότηση και δεν συμφωνώ με τη σχετική πρόταση γιατί πιστεύω ότι έτσι θα αποδυναμωθεί η γνωμοδότηση και νομίζω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να αποστείλει στην Επιτροπή Ανάπτυξης ένα ισχυρό μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο? Όχι. Έχουμε ολοκληρώσει το, το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. το οποίο θα ψηφίσουμε σε λιγάκι. Πάμε στο σημείο 6. Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών. Η κυρία Μάκιντάιρ. Συμφωνείτε να αρχίσουμε από την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα και μετά να πάρετε εσείς το λόγο. Συμφωνείτε? Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση να εξετάσουμε πρώτα την προφορική ερώτηση του σημείου 7 που είναι μία ερώτηση στην οποία καταλήξαμε στο περιθώριο των εργασιών της Επιτροπής Ήτρε για να είμαστε βέβαιοι ότι λαμβάνονται υπόψη επαρκώς τα ε, κοινωνικά ζητήματα και τα ζητήματα απασχόλησης. Οι συζητήσεις ε, επικεντρώθηκαν κυρίως ε, στις δομές ε, που δίνουν τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε δομές κοινωνικού διαλόγου. Κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελα να μην είναι πολύ δεσμευτικό αυτό το τμήμα και νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μία διατύπωση που να μπορεί να βρει όλους σας σύμφωνους ε, και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο για την προφορική αυτή, αυτή ερώτηση? Αν, ε, αν όχι, θα την ψηφίσουμε αργότερα. Στο μεταξύ όμως, να συζητήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες για το ψήφισμα. Πρώτον, μία νομική αναφορά που δεν δημιούργησε ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία αφορά το πώς θα ε, συνδυάσουμε το επαρκές επίπεδο των μισθών και από την άλλη τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την ασφάλεια όσον αφορά τη συμβιβαστική τροπολογία C. Ε, Για την παράγραφο 4 μιλάω. Υπήρξαν ε, αρκετές τροπολογίες ε, που έπρεπε να τις λάβουμε υπόψη. Σε σχέση δηλαδή με το τι ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις εθνικές δοκιμές. υποθέτω υπό το πνεύμα του σεβασμού ε, της ε, επικουρικότητας ε, θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εισβάλλει πάρα πολύ στην νομοθεσία των κρατών μελών. Θα παροτρύνει μεν αυτές τις εθνικές δοκιμές, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τον ορισμό ε, συστηματικών προτύπων ε, τα οποία να πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά τώρα το σημείο D, τρεις ε, συνάδελφοι συμφωνούσαν επ' αυτού και αναφερόταν στη σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την η ανησυχία αυτή αφορούσε κυρίως το υπερβολικό γραφοκρατικό άχθος για τις επιχειρήσεις και από την άλλη έπρεπε να υπάρχουν συστάσεις, ε, υπάρχουν και οι συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Προσπαθήσαμε να υπάρχει ένα ε, σε ευρωπαϊκός για το θέμα αυτό. Τα μαγειρέψαμε κάπως για να το πω έτσι αλλά από τη μία προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη του στόχου τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία και από την άλλη έχουμε λάβει υπόψη την ανησυχία του Φιλίπ Μπουλό ο οποίος ε, ούτω ή άλλως ε, ως εισηγητή ε, για τον προπολογισμό, ήθελε να τονίσουμε ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα. Όσον αφορά τώρα το πέμπτο, τον πέμπτο συμβιβασμό, αφορούσε, αφορά το κατά πόσο συστηματικά ή όχι, πώς περικόπτουμε το γραφειοκρατικό άχθος και νομίζω ότι έχουμε βρει μια αρκετά καλή ισορροπία, υπενθυμίζοντας ε, το ρόλο των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και την προστασία των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έκτος και τελευταίος συμβιβασμός ε, και πάλι καταφέραμε να συγκεράσουμε τις απόψεις των συναδέλφων πολλών ομάδων για να ε, συνδυάσουμε το επίπεδο της συμμετοχής σε αυτές τις δομές πρέπει όντως να υπάρχει, αλλά να ε, υπενθυμίζουμε και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Θέλει κανείς από όσους υπέβαλαν τροπολογίες να πάρουν το λόγο ή κάποιος άλλος συνάδελφος. Αν όχι, να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Θα, θα το ψηφίσουμε αυτό το θέμα ε, στη συνέχεια. Α, ναι, κύρια Γιαζουβιέτσκα, βεβαίως. Να σας δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση για την τροπολογία 4. Τι εννοείται με την προαγωγή των διτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Και στην τροπολογία 6 βλέπω μία δήλωση ότι οι γυναίκες που ε, ε, εργάζονται κατά μόνας δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό αποτυχίας ή βαθμό αποτυχίας όπως οι άντρες. Πώς ε, καταλήγετε σε αυτά τα συμπεράσματα. Sur, euh, Madame, c'est sur quel euh, για ποια παράγραφο ακριβώς ε, ομιλείτε. Τροπολογία 4, Στάκενμπουργκ και 6, Χίρσ. Τροπολογία 6. Στην 4 βλέπουμε την εξή δήλωση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξη της διάδοσης της εναλλασσόμενης κατάρτισης ε, στα ελληνικά ε, και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Και στην τροπολογία 6 της κυρίας Νάντια Χίρς βλέπω την εξή δήλωση. Οι γυναίκες που αποφασίσουν να αρχίσουν δική τους επαγγελματική ε, δραστηριότητα δεν αποτυγχάνουν στον ίδιο βαθμό όπως οι άντρες. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, κάποιες έρευνες ε, να μας παραπέμψετε. Euh, Κυρία Μάκιντιρ. Ήθελα να ευχαριστήσω για τις συμβιβαστικές τροπολογίες εκτός από αυτές που έχουν συμπεριληφθεί. Το ECR είναι υπέρ της E και της F συμβιβαστικών τροπολογιών. Ήθελα αυτό να προσθεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Ο κύριος Μπινιού. Ναι. Μας πήραν χρόνο οι συμβιβαστικέ, αλλά γενικά είναι καλές. Είναι ευρείες, ευρείς συμβιβασμοί, διαπαραταξιακά, που εκφράζονται μέσα, το, μέσα από τις τροπολογίες. Με την ΆΗ δεν συμφωνώ, γιατί αφαιρέθηκαν πράγματα έτσι που τα θέλαμε, χωρίς να προσθεθεί κάτι από αυτά που θέλαμε να προσθεθούν. Οπότε προτιμούμε το αρχικό κείμενο σε σχέση με τη συμβιβαστική ΆΗ. Η, η κυρία Μακίνταερ χωρίς μικρόφωνο. Α, είμαστε στην προφορική. Η κυρία Μακιντάιρ, νομίζω ότι το ερώτημα της ε, συναδέλφου για την τροπολογία 6 ήταν στη δική μου και όχι στη δική σας έκθεση. Οπότε, ναι, νόμισα ότι συζητούσαμε τη δική σας. Ναι, άλλαξα την ημερήσια διάταξη, ενώ δεν έπρεπε, χωρίς να το πω. Δεν ενημέρωσα κανονικά. Συγγνώμη για τη σύγχυση. Τώρα συζητάμε την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα μετά την έκθεση της κυρίας Μακιντάιρ που αφορά την ε, ανασκόπηση των ΜΜΕ από την Επιτροπή. Ναι, αλλά για την ε, προφορική ερώτηση αφορά όλες τις ε, συμβιβαστικές. Εγώ πάντως νόμιζα ότι επειδή μιλούσαμε για την τροπολογία 6 είχαμε προχωρήσει. Επιστρέφω στη γλώσσα του Φρανσουά Ολόντ. Συμπεραίνω ότι δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο και άρα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα και στη συνέχεια θα το ψηφίσουμε. Αλλά πριν ψηφίσουμε έχουμε ακόμη δύο σημεία να εξετάσουμε. Πρώτον, την εξέταση, πρώτον την ε, έκθεση της κυρίας Μάκιντάρ και των συμβιβαστικών τροπολογιών. Η κυρία Γιαζουβιέσκα ήδη πήρε το λόγο για το θέμα αυτό, αλλά πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Μάκιντάιρ για να μας εξηγήσει περισσότερο και λεπτομερέστερα τις συμβιβαστικές τροπολογίες της εκθεσής της, ε, που είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις ε, εμπορικές προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους τους κοιόδης για τη συμβολή και τη μεγάλη συνεργασία και χαίρομαι που μπορέσαμε να φτάσουμε σε τόσο πολλές συμβιβαστικές. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή παρενέβαινε και έκανε τις αλλαγές και εκτίμησα πολύ το έργο τους. Θα αποσύρω τις 44 και 60 τροπολογίες μου, σας το λέω ε, παρόλο που το είχαμε κοινοποιήσει. Αυτές οι δύο τροπολογίες θα αποσυρθούν. Και πιστεύω ότι η κυρία Ρέτνερ θα αποσύρει την 1 και 2, που πολύ το εκτιμώ αυτό. Να σας πω για το λόγο. Δεν είναι ότι διαφωνούμε με τις τροπολογίες, αλλά στη γνωμοδότηση δεν υπάρχουν ε, παράγραφοι που να είναι σαν αιτιολογικές σκέψεις ε, και θέλαμε να υπάρχει σωστή ισορροπία, να είναι ισορροπημένη η έκθεση. Αν αποσυρθούν αυτό θα είναι καλό. Αρχίσαμε με 62 τροπολογίες και τελειώσαμε με 12 συμβιβαστικές και γενικά όλοι συμφωνούν με τους συνολικούς στόχους και προτάσεις. Το καλό που ε, με το γεγονός ότι αρχίσαμε με γνωμοδότηση είναι ότι είναι μικρό το κείμενο αρχικά και μπορούσαμε να το επεκτείνουμε με παραγράφους, να προσθέσουμε και να συμπεριλάβουμε πράγματα που είναι σημαντικά για τις ε, ομάδες, τις πολιτικές ομάδες. Γενικά δεν πιστεύω ότι το σημείο εκκινήσεως άλλαξε αλλά έχουν προσθεθεί σημεία. Ειδικότερα φροντίσαμε να συμπεριληφθεί η υγεία και η υγιεινή και η ασφάλεια, να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο χωρίς να ε, διακινδυνεύσουν άνθρωποι, χωρίς να τους βάλουμε σε κίνδυνο. Πολύ το θέλαμε αυτό το σημείο. Επίσης, ε, ειδική μνήμα για τις γυναίκες επιχειρηματίες υπάρχει. Και μάλιστα για να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με την τροπολογία 6, προσθέσαμε ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά δεν συμπεριλάβαμε την μάλλον η πιθανόν υποκειμενική άποψη ότι οι γυναίκες δεν αποτυγχάνουν τόσο συχνά όσο οι άνδρες. Τα άλλα τα συμπεριλάβαμε. Ε, και για την κυρία Σρότερ που ανησυχούσε συμπεριλάβαμε και την ιδέα των διασυνοριακών υπηρεσιών και των μόνο απευθυντικών θηρίδων και πιστεύω ότι αυ... και ξέρω ότι αυτό την απασχολούσε ιδιαίτερα. Ξέρω ότι μπορεί μας είχαν ειδοποιήσει ότι ο κύριος Σπάνιον δεν θα ε, συμφωνούσε με μια συμβιβαστική, αλλά είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι είχαμε ευρεία διαπαραταξιακή συνεργασία και οι περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες υποστηρίζονται από όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ όλους λοιπόν για την δουλειά αυτή που έκαναν. Ευχαριστώ. Κυρία Γιαζιοβιέτσκα. Η κυρία Σρότερ και η κυρία Στάινρουκ ε, είχαν, είχαν υποβάλει τροπολογίες και η κυρία Χίρς. Κυρία ε, Ρέγνερ, θέλετε να απαντήσετε. Ε, με δύο λόγια υποστηρίζω και τονίζω αυτό που είπε και η κυρία Μάκιντάιρ στις διαπραγματεύσεις μας ως κοιόδης στην αρχή ξεκινήσαμε από διαφορετικές θέσεις. Από τη μια πλευρά ήταν η μεγάλη προτεραιότητα ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει πάντοτε να ελαφρυνθούν και να απελευθερωθούν από γραφειοκρατικά εμπόδια και από την άλλη πλευρά υπήρχε ο μεγάλος μου φόβος να μπερδέψουμε ανώμια μεγέθη ε, θέματα υγιεινής, προστασίας των εργαζομένων κλπ. Και πράγματι καταφέραμε αυτές τις ε, παρανοήσεις όχι μόνο να τις ε, εξαλείψουμε αλλά να ε, βρούμε κοινούς στόχους που αντικατοπτρίζονται στις συμβιβαστικές. Θέλουμε όλοι να διευκολύνουμε τη ζωή των ΜΜΕ για να έχουν επιτυχίες, να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία και από την άλλη πλευρά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και είναι σαν κόκκινη κλωστή στο κείμενό μας, να φροντίσουμε ότι θα είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για golden plating όταν μιλάμε για ασφάλεια των εργαζομένων, ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά πρόκειται για ελάχιστα πρότυπα και ότι ε, αυτά δεν θα πρέπει να ε, είναι σε αντίφαση μεταξύ τους. Γι' αυτό η διατύπωση των συμβιβαστικών τροπολογιών βέβαια δημιουργήθηκαν την τελευταία στιγμή, αλλά όλοι ε, είχαμε ένα πνεύμα ε, επικοδομητικής ε, συνεργασίας και βούλησης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Κυρία Γιαζιοβιέτσκα κυρία Πρόεδρε. Είχα ζητήσει κάποιες εξηγήσεις και για την ε, συμβαστική α και την τροπολογία 4. Αυτή την, ε, αφορά στην διάδοση της εναλλασσόμενης κατάρτισης. Δεν κατανοώ τον όρο εναλλασσόμενη κατάρτιση. Θα ήθελε κανείς να μου το εξηγήσει. Bei der dualen Berufsausbildung είναι το διαδικό σύστημα που έχουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ επιτυχημένο στην Ευρώπη. Μετά το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης υπάρχει δυνατότητα παράλληλα σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και σε θέσεις μαθητείας σε έναν εργοδότη, σε μια επιχείρηση, μπορεί κανείς να μάθει ένα επάγγελμα. Αυτό είναι το λεγόμενο διαδικό σύστημα, το οποίο έχει καταξιωθεί στη Γερμανία, την Αυστρία και σε τροποποιημένη μορφή και στην Ολλανδία, για παράδειγμα. Ε, και χαρακτηρίζεται από την πρακτική άσκηση, είναι κοντά στην πράξη. Δηλαδή, ε, βλέπουν ποιες ανάγκες υπάρχουν στις επιχειρήσεις και εκπαιδεύουν, καταρτίζουν αντίστοιχα τους νέους ανθρώπους. Οι χώρες που έχουν αυτό το λεγόμενο διαδικό ή εναλλασσόμενο, όπως λέμε, σύστημα, έχουν την λιγότερη, κατά πολύ λιγότερη ανεργία των νέων, γιατί ε, μπορεί κανείς ε, με ήπιο τρόπο να προσαρμοστεί στις ανάγκες της οικονομίας και του, του κόσμου της εργασίας και οι νέοι βρίσκουν ε, θέση. Και ο, πρόεδρο ο πρόεδρος της Επιτροπής Μαρόζο, αλλά και άλλοι εξετάζουν πώς αυτές οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να εξαπλωθούν πάντοτε προφανώς λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Γιατί προφανώς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, αλλά θέλουμε να ε, αναδείξουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τα θετικά στοιχεία από αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσει και Ζουβέτσκα. Ναι, βεβαίω είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την απάντηση. Με καλύπτει. Κατανοώ λοιπόν ε, θεωρητικά ε, αυτό το σύστημα, το διαδικό σύστημα κατάρτισης. Ε, με προβλημάτιζε ο όρος. Οι εξηγήσει μας ήταν πολύ σαφεί. Ευχαριστώ θερμά. Παρόμοια συστήματα βεβαίω υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ίσως ο όρος ήταν αυτός που με μπέρδεψε. Ευχαριστώ. Parfait. Tout l'importance parfois des débats en commission. Πολύ ωραία. Αυτές οι συζητήσεις ακριβώς είναι στην Επιτροπή μας που δίνουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε ε, το εθνικό επίπεδο κατανόησης, ε, κατανόησής μας. Κυρία Μακίνταϊρ, θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο? Όχι. Ωραία. Δέκα η ώρα θα ψηφίσουμε. Έτσι είχαμε ενημερώσει άλλωστε και τα μέλη της Επιτροπής ότι θα ψηφίζαμε στις 10. Μας έχουν μείνει όμως 10 λεπτάκια. Οπότε θα υποφεληθώ για να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης του οποίου εγώ ε, είμαι υπεύθυνη για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρόκειται για μία γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών βεβαίως ε, και αποτελεί τμήμα της οριζόντιας διαδικασίας στην οποία συμμετέχει και η δική μας Επιτροπή. Γνωρίζετε άλλωστε και την έκθεση κόζας για το γενικό ε, κανονισμό ε, της κυρίας Ζατιέ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της κυρίας Στάινρουκ για το Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρόγραμμα και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Σε αυτή τη γνωμοδότηση προτείνω καταρχάς κάποια στοιχεία πραγματολογικά για να υπενθυμίσω τι ακριβώς ε, σημαίνει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι κοινωνικές πτυχές ε, και λόγω των ε, ανισοτήτων που υπάρχουν των μακροοικονομικών και για να μπορέσουμε να έχουμε μία αντικυκλική πολιτική και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την αποφάσισε στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα θυμάστε ότι επί των πέντε στόχων Στου στους οποίους αποφασίσαμε. Ε, τρεις έχουν να κάνουν με τη δική μας ε, ε, αρμοδιότητα, δηλαδή μια καλή κοινωνική πολιτική. Και όταν συζητούμε τέτοιου είδους θέματα βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε και μία σημαντική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την μακροοικονομική επιλεξιμότητα προτείνω να μην ε, την ε, ε, διατηρήσουμε ως στοιχείο γιατί χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ βέβαια των περιφερειών και των τοπικών αρχών. Επίσης θα, θέλουμε, θα θέλαμε να επιμείνουμε για τη σημασία των κοινωνικών πολιτικών προκειμένου να υπάρξουν πολιτικές που θα ανταποκριθούν στις ε, διαρθρωτικές προκλήσεις ε, που έχουν να κάνουν είτε με την ανεργία ε, μεγάλης διάρκειας και νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία δεν είχαν απασχολήσει ούτε τον νομοθέτη ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα και μιλάω για το άρθρο 9 που θα έπρεπε να είναι ε, το επίκεντρο της σχετικής νομοθεσίας. Θα ήθελα να επιμείνουμε επίσης όσον αφορά στα ποσοστά. Νομίζω ότι είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα ε, την Επιτροπή μας. Ε, στην, κυρία, στην έκθεση της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ φάνηκε αυτό να επιμείνουμε στο 25% του ΕΚΤ και στο 20% για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την ε, κοινωνική ένταξη. Νομίζω ότι τροποποιήσαμε και τον τίτλο για να συμπεριλαμβάνεται η μη διάκριση. Από αυτό παρεκκλίνουμε βέβαια, με αυτό παρεκκλίνουμε σε σχέση με αυτό που ψηφίσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να το επανεπισημάνουμε αυτό και είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει επίσης ε, η επανεπισήμανση της υποστήριξης ε, των κρατών μελών όταν αυτό χρειάζεται και τους επιτόπου φορείς όσον αφορά τις ε, διοικητικές ικανότητες, τις διοικητικές δομές, γιατί είναι γεγονός ότι τα κονδύλια του ΕΚΤ, των Ευρωπαϊκών Ταμείων, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να υποκαθιστούν την εθνική ε, διοίκηση. Παράλληλα βλέπουμε ότι όταν αξιοποιούνται σωστά τα κονδύλια, πρόκειται για χώρες στις οποίες ε, η διοικητική ε, δραστηριότητα είναι κάτι το παραδοσιακό και εκπονείται με ιδιαίτερο επαγγελματισμό. Αν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, τα κράτη κατηγορούνται για υποαξιοποίηση των κονδυλίων, για διαφθορά και εμείς βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ε, ε, διοικητική διαχείριση. Να ξαναπούμε δηλαδή αυτό που είχαμε πει και στην έκθεση Steinruck για την αναγκαιότητα συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών. Η τέταρτη πτυχή επίσης και η σχετική συνεργασία για τους νέους μιλούμε με ε, την τροποποίηση βέβαια του ε, δημοσιονομικού ε, σκέλους που έχει να κάνει με αυτό το θέμα και την αύξηση των ποσοστών. Στην πρώτη έκθεση της κυρίας Άρκιν για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας από τους γενικούς προσανατολισμούς προσέγγισης έκθεσης αυτής που λέει ότι περνάμε ε, στο Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης σε μια ευρύτερη προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπιστεί το θέμα της αναδιάρθρωσης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη γνωμοδότηση να, επισημάνουμε εκ νέου την δέσμευσή μας να υπάρχει ένα πρόγραμμα επισητιστικής, βοήθεια, βοήθειας για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Ξέρετε την ε, ε, τρομερά κακή δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε ότι οι φτωχότερες χώρες ε, έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα με τρομερές ανεπάρκειες και αδυναμίες. Υπάρχουν σοβαρές επιστητιστικές αδυναμίες και Θέλουμε στο πλαίσιο της επικουρικότητας να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα στις χώρες αυτές για να τις βοηθήσουμε και το οποίο βέβαια συνάδει με την ε, ευρύτερη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητούμε τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από το δικό μας ψήφισμα υποσχέθηκε στην Ολομέλεια να επανέλθει με μια πρόταση για το θέμα αυτό. Από ό,τι κατάλαβα θα το κάνει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να συζητήσουμε αυτή την νομοθετική βάση, τη νέα νομοθετική βάση, να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και παράλληλα το σημείο της απασχόλησης να ληφθεί υπόψη σοβαρά στο πλαίσιο των πολιετών δημοσιονομικών ε, προοπτικών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και για μένα Γι' αυτό σα εξηγώ για ποιο λόγο πρέπει να, να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα. Εξού και η πρότασή μου. Ξέρω ότι η κυρία Σρότερ δεν συμφωνεί με αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τις επιτροπές παρακολούθησης και κατά πόσο οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν ώστε να συμμετέχουν περισσότερο οι επιτόπου φορείς και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Νομίζω ότι ο ρόλος του νομοθέτη δεν είναι να είναι κανείς ε, στο συνεφάκι του. Ε, εμείς είμαστε οι καλύτεροι υπέρμαχοι αυτών των προγραμμάτων, αυτών των προσανατολισμών και θέλουμε να υπάρχει και ένα πολιτικός, ε, να υπάρχει ένας πολιτικός ευανάγνωστος χαρακτήρας, ορατός χαρακτήρας. Εξού και οι επιτροπές αυτές παρακολούθησης υπάρχει μια υποχρέωση χρέωση παρακολούθηση από πλευρά μας. Ε, η κυρία Σρότερ τα ξέρει όλα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γνωρίζει όλα τα προγράμματα των ε, διαφόρων κρατών μελών ε, και φαντάζομαι κυρίως της Γερμανίας, αλλά όταν σκεφτόμαστε για παράδειγμα τη χρηστή διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, είναι μια πρόταση νομίζω που χρήζει επεξεργασίας ε, και συνέχισή. και νομίζω ότι βάσει αυτής της πρότασης μπορούμε να φτάσουμε όλοι μαζί σε μια συμφωνία. Και τέλος, δεδομένου βέβαια του, δεδομένης της για τον προπολογισμό, Πρέπει να πούμε και κάτι για τους ε, οργανισμούς, τις υπηρεσίες, γιατί ξέρουμε ότι είναι σημαντικό για τις δικές μας, για δικά μας καθήκοντα, αν θέλουμε να εισακουστεί η φωνή μας ε, ε, σε σχέση με τα άλλα επιχειρήματα που θα ακουστούν υπέρ της δημοσιονομικής διαιτησίας. Σας τα είπα κάπως φορτωμένα, αλλά είμαι υποχρεωμένη. Είμαι υποχρεωμένη να σας, αναφερθώ επίσης, να σας αναφέρω επίσης και μια τροπολογία που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει σε σχέση με τη διοργανική συμφωνία στο πλαίσιο της ε, συνεργασίας για τον προϋπολογισμό και έχει να κάνει με το μέλλον ε, της, ε, του, ταμείου, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, δεδομένων των γενικών προσανατολισμών που θέλουμε να δώσουμε στο συγκεκριμένο ταμείο. Ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Συγγνώμη, μακρηγόρησα, αλλά έτσι δεν θα διαβάσετε τη γνωμοδότηση. Και πιστεύω ότι έχετε στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Άρχεται η συζήτηση. Φαντάζομαι ότι δεν θα υποβάλλετε για τροπολογίε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλει και κανεί να πάρει το λόγο. Όχι. Ωραία. Τότε Αν το χάσατε μπορείτε ε, να ε, καλύψετε τα κενά σας ε, μέχρι τις 10 Ιουλίου 12 το μεσημέρι και να υποβάλλετε τροπολογίες. Αν όλα πάνε καλά, θα εξετάσουμε στις 6 Σεπτεμβρίου τις τροπολογίες, 17 και 18 την γνωμοδότηση, 17 την γνωμοδότηση και 18 να ψηφίσουμε. Φτάνουμε λοιπόν στην ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Je vous propose euh, Καλύτερα να ψηφίσουμε πρώτα το 12 που είναι η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Και κάτι άλλο. Είχε σωτμά κι άλλα εδώ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, ένα αίτημα να απευθύνω. Μπορούμε παρακαλώ να ψηφίσουμε με τη σειρά του καταλόγου ψηφοφορίας. Ήταν μια ιδέα τη τελευταία ε, στιγμή, αλλά θα τα ξαναπώ για να είμαστε σαφεί. Θα ψηφίσουμε κατόπιν τη κυρία Μακίντάιρ ε, τις εκθέσεις όπως είχαν προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη αρχικά. Δηλαδή πρώτα το, ψηφίο, το σημείο 11 Το σχέδιο γνωμοδότησης τη κυρίας Μάκιντάρ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, Τροπολογία 1, Ρέγνερ, έχει αποσυρθεί, όπως και οι δύο. Έχουμε συμβιβαστική τροπολογία Α από 5 ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συμβιβαστική B από 5, από ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 σρόντερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 σρόντερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 ε, συμβιβαστική τροπολογία από τέσσερις ομάδες ε, εργασίας. Σωστά κυρία με κάντε. Ωραία. Σι λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέντε ομάδες τελικά είχαν υποβάλει τη συμβαστική αυτή. Λοιπόν, μένουμε στην παράγραφο 3, δεύτερη συμβιβαστική ή πέντε ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κυρία Ρέγνερ. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, για τη συμβαστική D. Εκεί θέλω να υποβάλω προφορική τροπολογία όταν φτάσετε, Πρόεδρε. Το συζητήσαμε με την εισηγήτρια. Αντί για, το... Ε, αντί για συχνά να πούμε ότι δύναται σε αυτή την τροπολογία. Can you tell me a bit more about it because I don't Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε καλύτερα γιατί δεν το βρίσκω στο κείμενο. Γιατί μείωση του διοικητικού άκου δεν θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας της υγείας για τους εργαζομένους. Γιατί συχνά αυτό το άχθος οδηγεί σε α, στρες Μπορείτε, α, can result στα αγγλικά. Μπορεί, δύναται να οδηγήσει. Can result να φύγει το often στα αγγλικά, το συχνά. Um, Μάλιστα. Επί της βάσης αυτής, μετά την παράγραφο 3, ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική D με την προφορική τροπολογία. Δεν διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική D όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι πράσινοι καταψήφισαν. Λοιπόν, τροπολογία 21. Υπέρ της 21. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Πολ Μάρφη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 καταπίπτει, οπότε ψηφίζουμε την 24 του Πολ Μόρφη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 καταπίπτει, την 26 ψηφίζουμε. Του κυρίου Πουπάκη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 27 της κυρίας Σρόντερ. Δύο τμήματα. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε την 28. Μάκινταρ. Υπέρ της 28. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. 29 καταπίπτει αν εγκριθεί 23, αλλά 23 κατέπεσε. Άρα καταπέπτει και αυτή. Άρα, μετά πάμε στην τροπολογία 30 παράγραφος 4. Νικόλ Μανέσκου, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F τριών ομάδων. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 34 με προφορική τροπολογία της ECR. Διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία? Όχι, οπότε την ψηφίζουμε. Όπως τροποποιήθηκε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά, να την ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Ψηφίζουμε τη 34 ηλεκτρονικώς άρχια ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21-14 εγκρίνεται σαφέστατα. Τροπολογία 33 Ρέγνερ Στάινρουκ. Συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμφωνούμε. Ωραία. Τροπολογία 35 καταπίπτει. Οπότε, παράγραφος 5 καταπίπτουν οι σχετικές τροπολογίες και περνάμε στη συμβιβαστική G για την παράγραφο 6 εκ μέρους τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική K. Από τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 44, έχει αποσυρθεί, οπότε πάμε στην παράγραφο 7, συμβιβαστική H, εκ μέρους τριών ομάδων υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται συμβιβαστική L, από τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία I εκ μέρους δύο ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 Ρέγνερ και Στάινρουκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 Σρέντερ υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Φύσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 19-16. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 συμβιβαστική Jake μέρους 4 ομάδων υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 Μπέκερ υπέρ. Κατά. Υπέρ και πάλι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 έχει αποσυρθεί. Μετά, παράγραφος 9, 61, χίρς, δύο τμήματα, γιατί έτσι ζήτησε ECR. Ψηφίζουμε το σύνολο εκτός από το While Still Maintaining the European Social Model, υπέρ της 61, χωρίς, αυτά τα, χωρίς αυτή τη φράση, κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ευτυχώς. Τροπολογία 54 στην παράγραφο 8 της κυρίας Σρέντερ καταπίπτει γιατί έχει καλυφθεί από τη συμβιβαστική L. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της ε, γνωμοδότησης ε, ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία μας, το σημείο 12. Πρώτα την προφορική ερώτηση για την ελαχιστοποίηση ρυθμιστικού φόρτου για τις μικρομισές επιχειρήσεις. Για, το ερω... για την ερώτηση 1, τροπολογία 2 του Φιλ Μπενιόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Σρόντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, μετά την ερώτηση, μετά, σε δύο τμήματα και υπάρχει και προφορική τροπολογία. Για το πρώτο τμήμα, ένα λεπτό, ένα λεπτό λέει η Πρόεδρος. Πρώτο τμήμα, would the Commission agree μέχρι EU legislation in the field of employment law is respected. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Και η προφορική τροπολογία που σας προτείνω είναι να διαγραφεί το relatively. Κύριε Ουρή, θέλετε να πάρετε το λόγο. Η προφορική τροπολογία 3 έχει καταπέσει. Η τροπολογία 3 έχει καταπέσει. Και εγώ βλέπω στον κατάλογό μου ότι η 1 καταπίπτει εάν εγκριθεί η 3. Δεν ψηφίσαμε όμως εμείς την 1. Πρόεδρος, μπορεί να μην έχουμε τον ίδιο κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά εγώ βλέπω στο σχόλιο για την 1 ότι καταπίπτει αν η 2 εγκριθεί και ότι είναι συμβατή με την 3. Επειδή όμως κατέπεσε με την τροπολογία 2 που ψηφίσαμε, άρα δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε πλέον. Γιατί ψηφίσαμε τη 2, κατέπεσε και συνεπώς δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Γιατί έτσι είναι η ιεράρχηση της, ε, του, του καταλόγου της ψηφοφορίας. Πρώτα βλέπουμε αν καταπίπτει και μετά αν είναι συμβατή. Επανερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 4 της κυρίας Μάκιντάιρ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίζουμε τώρα το υπόλοιπο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά το, την ερώτηση 1, τροπολογία 5 Σρέντερ πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, μάλλον το, το σύνολο του κειμένου εκτός, αυτό, εκτός από το with particular attention transnational services provision. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, how will the commission ensure EOS standards in the single market. Αυτό το τμήμα ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ της συμπερίληψης, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ερώτηση 2. Συμβιβαστική α εκ μέρους τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε τώρα την 9 Μάκιντάιρ υπέρ κατά Α, δεν ψηφίζετε πια. εννιά και πάλι, υπέρ. Για την εννιά μιλάω. Υπέρ. Τροπολογία 9 υπέρ, επαναλαμβάνω. Κατά. Λοιπόν, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός ε, γιατί βλέπω ότι τα έχουμε χάσει λίγο. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για να είμαστε σίγουροι. Για την τροπολογία 9. Ψηφίσατε όλοι. Οπότε, πέρασε τη ψηφοφορία. 24 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. Η τροπολογία νέα της κυρίας Μάκιντάρ εγκρίνεται επομένως. Οπότε, φτάνουμε στην ερώτηση 4, τροπολογία 10 Μάκιντάρ. Είναι κατά η συγγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Εντάξει, να ελέγξουμε τροπολογία 10. Έναρξη ψηφοφορίας. Alors, euh, le vote est Πέρα της ψηφοφορίας. Συγγνώμη, είναι πολύ αργά. Είναι η απάντηση σε μια ερώτηση που δεν ακούσαμε γιατί ήταν εκτό μικροφώνου. 34 κάρτε. 36 ψήφισαν, 6 ε, υπέρ, 30 κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται τι λέτε εσείς. Οπότε επιβεβαιώνεται η ψηφοφορία που κάναμε προηγουμένως. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Ah, c'est Πέρα τη ψηφοφορία τη ηλεκτρονική, ε, οπότε Εγκρίνεται η προφορική ερώτηση, 35 υπέρ, 0 κατά και 2 αποχές. Για να μην έχετε την εντύπωση ότι η συγγήτριά σας ε, ήταν πλήρως αναποφάσιστη, θα σας ε, εξηγήσω τι έγινε με την τροπολογία 9 της ε, κυρίας Μακεντάιρ. Κάνω κατάχρηση της θέσης μου ως Προέδρου θελήσαμε να αποσυρθεί από τα πρακτικά αυτή η ψηφοφορία γιατί ήταν μια γλωσσική τροπολογία για την οποία δεν θα έπρεπε να ψηφίσουμε. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν είχατε καμία ένδειξη ε, της ε, ε, θέσης της συγγήτριας. Φτάνουμε τώρα στο νομοθέτημα. Τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 Μάκιντα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 6 Κρόιτσμαν υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 7 Μπινιόν υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται παράγραφος 3 συμβιβαστική B εκ μέρους 6 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία για την οποία δεν διαφωνεί κανείς, οπότε ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 συμβιβαστική C εκ μέρους τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε σε διαφωνείτε με τη συμβιβαστική ΣΥ. Μάλιστα. Μάλλον επειδή δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας μου, λέει εκτός μικροφώνου ο κύριος Κρίστενσεν. Ψηφίσαμε τη συμβιβαστική ΣΥ. Ξέχασα να το πω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε με μια προφορική τροπολογία για να μην υπάρχει το however στο κείμενο το, είχε ζητήσει αυτό, το είχαν ζητήσει φιλελεύθεροι. Λοιπόν, παράγραφος 5, τροπολογία 14, McIntyre. Για διαγραφή, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, Κρόιτσμαν Μπένιον, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 15 του Μπένιον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 Νταρντέν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 18 καταπίπτει, άρα παράγραφος 6, τροπολογία 20, μπενιών με προφορική τροπολογία. το lowering να, να ε, τροποποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί το adaptation. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, Christensen Ludwigson, δύο τμήματα. Το σύνολο του κειμένου χωρίς το offering financial incentives, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ της προσθήκης του κειμένου, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 7, δύο τροπολογίες διαγραφής, 22 του Κρόιτσμαν και 23 Μάκιντάρ. Είναι ταυτόσημες. ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική τροπολογία D εκ μέρου τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολόγια 28, Ταρντέν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολόγια 29, Κρόιτσμαν, Μπένιον, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Κυρία, Μαρ... Κυρία Αρκίν, διαφωνείτε με την ε, τροπολογία του κυρίου Κρόιτσμαν. Μάλιστα. Ίσως να πήγα πολύ γρήγορα. Τροπολογία 30 Μάκινταρ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 Φιλίπ Μπουλόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 συμβιβαστική ε, Ή από 4 ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 συμβιβαστική τροπολογία F εκ μέρους Τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 τροπολογία 40 Κρόιτσμαν και Μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 Μπουλόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 42 τροπολογία Σρόντερ με προφορική τροπολογία διαγραφή του End of Enterprises of the Social Economy. Υπέρ τη 42 όπως τροποποιήθηκε, κατά, αποχές, καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, ωραία. 21-17, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 43, Κρόιτσμαν Μπένιον. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 44, Σρόντερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 15, τροπολογία 45-46, ταυτόσημες, για διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 47, ορί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16, Ψηφίσαμε στην παράγραφο 15 την τροπολογία 47 του κυρίου Τσάμπα Ορί. Η συγγήτρια... Ε, τι είπα εγώ. Α, συγγνώμη, έκανα λάθο, λέει η πρόεδρο. Γιατί είπα ότι το 45 και το 46 είναι. Ότι 45, 45 και 46 είναι ταυτόσιμε. Λάθο έκανα. Λάθο έκανα. Να ψηφίσουμε τη 46 Μάκιντα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα να μην ψηφίσουμε και πάλι τη 47, γιατί ούτως ή άλλως... Ε, α, καταπίπτει αν το 46 εγκριθεί. Αλλά η 46 Η 46 απορρίφθηκε, άρα πρέπει να ψηφίσουμε τη 47. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε τη 47 που την είχαμε ψηφίσει και πριν. Να την ξαναψηφίσουμε τη 47. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 47 του κυρίου Τσάμπα Ορή με θέση, με θέση υπέρ της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Πάμε στην παράγραφο 16, τροπολογία 48, Μάκινταρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Κρόιτσμαν, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική τροπολογία α στο... στην αιτιολογική σκέψη I. Πέντε ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 Schröder υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 36 υπέρ, κανεί κατά και δύο αποχές. Ευχαριστώ πολύ ο Πάμε στο σημείο 8 τώρα. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της Ντανούτα Γιαζιοβιέτσκα για το ε, Σύμφωνο Κοινωνικής Επένδυσης. Παράγραφος 1. Συμβιβαστική I. Εκ μέρους πέντε ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, il y a une faute sur ma liste de vote. Υπάρχει ένα σφάλμα στον κατάλογο ψηφοφορίας μου, φαντάζομαι το ίδιο και στο δικό σας κατάλογο, γιατί λέει εδώ ότι καταπίπτει αν η συμβιβαστική ε εγκριθεί, αλλά πρόκειται τελικά για τη συμβιβαστική I που μόλις ψηφίσαμε. Άρα, οι 46 και οι 47 λεπρόδος καταπίπτουν. Άρα μετά από την παράγραφο 1 μπορούμε να, ψηφι... μετά μπορούμε να ψηφίσουμε την 48 της ΕΣΑΙΑ, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της προστίκης, υπέρ κατά αποχές και πάλι εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 49 ΕΣΑΙΑ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 Μπερμάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 Στάινρουκ. Ε, συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Να ψηφίσουμε την 50. Να ψηφίσουμε και πάλι την 50 ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. 28 υπέρ 10 κατά. Κάτι άλλαξε και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 51 μπακ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβιβαστική J. Εκ μέρους πεντομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 58, Μάνερ και Χάρκιν. Με προφορική τροπολογία για τη διαγραφή της λέξης «κι», υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Συμβαστική και για την παράγραφο 4, από τρεις ομάδες, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 66 κάρμπνοχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για τον υπότιτλο τροπολογία 67 τούρουνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 σημείο A. Καλά, να ψηφίσουμε και πάλι την 67 ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ 21 κατά καμία αποχή. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική L. 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 72 του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές. Ξανά υπέρ της 72. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική M. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, τώρα πάμε στην 72 του Ρούνεν. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε, ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. σημείο B, συμβιβαστική N, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 εσάια, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο C, τροπολογία 81, μπουλόν. καταπίπτει γιατί έχουμε ψηφίσει με μια περίεργη αλφαβητική σειρά το, τη συμβιβαστική όμικρον. 85. Μπουλόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Βεβαίως κύριε Αντιπρόεδρε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό στην 85 πάντοτε θέλουμε να σας ευχαριστούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα που όλοι ψήφισαν, πέρα της ψηφοφορίας, 32 υπέρ και 2 κατά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαν. Τροπολογία 86 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 σημείο D 88 εσάια υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 87 της κυρίας Παπαδοπούλου. Συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σημείο Ι, e, συμβιβαστική π, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο σημείο F. Τροπολογία 97 μπουλόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 της κυρίας Εσάγια, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 α, τροπολογία 99 καταπίπτει, άρα πάμε στην παράγραφο 6, τη συμβιβαστική R, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, συμβιβαστική S. Πέντε ομάδες, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία γλωσσική που δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Όμως μετά την, τροπολογία 116 του κυρίου Κάμπρνοχ πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 8, συμβιβαστική τ. από 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 χείρους υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10 συμβιβαστική Β εκ μέρους 5 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Υπότιτλος 3, τροπολογία 137 εισαγια για διαγραφή υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 11, συμβιβαστική W, από 5 ομάδες υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 141 μπουλόν υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε την 141 του κυρίου Μπουλόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, 22-14. Αγκρίνεται. Πάμε λοιπόν την 140 ΕΣΑΓΙΑ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 142 Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 Ομπερμάιερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 13 συμβαστική X υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Πάμε τώρα παράγραφος 13, τροπολογία 148 του Ρούνεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Τροπολογία 149 εσάγια για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τότε την 151 κάμπρνοχ υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς γιατί δεν σηκώνται τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, 23-13 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Άρα, παράγραφος 15. 152 εισάγια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 ρέγνερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρο. Πρέπει να ψηφίσουμε την 154 τη κυρία Παπαδοπούλου. Ψηφίζουμε την 154 τη κυρία Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε. Εκτιμώντα τροπολογία 1, ε, Μάνερ και Χάρκιν υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Μετά τροπολογία 2, Γκέντς υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 γκόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 μάνερ και χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 κάμπρινοχ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική B. Τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C από πέντε ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 μπουλών Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 κυρία Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την τροπολογία 40 της κυρία Παπαδοπούλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18-15 και τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Μετά, τροπολογία 41 του Ρούνεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αν σηκώνετε το χεράκι καλύτερα θα είναι. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 Στάινρουκ υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε τη 42 της κυρίας Στάινρουκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 υπέρ, 18 κατά και μία αποχή. Δεν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 37 ψηφίσαντες, 35 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Κυρία Γιαζιουβιέτσκα. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Έμερ Κοστέλο για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 2011. Παράγραφος 3, συγγνώμη κύριε Μπουλό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποσύρω την ε, τροπολογία μου, την υπαριθμόν 1. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Δεν ψηφίζουμε γενικώ. Ψηφίζουμε τη 2 της κυρίας Μάνερ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα την 3 Λάμπερτ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην παράγραφο 4, τροπολογία 6, Φιλίπ Μπουλόν. Πέντε τμήματα. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου χωρίς το binding, obligations and και calls on the commission μέχρι το enforcement of these obligations. Ψηφίζουμε δηλαδή το πιο soft κομμάτι ας πούμε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ποιος θέλει binding. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν θα έχουμε το binding. Ποιος θέλει obligations end. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ποιος θέλει να προσθεθεί of encourage. Α, μέχρι το of encouraging employers μέχρι το social label. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ποιος είναι για το υπο, υπέρ του υπόλοιπου κειμένου, κατά, αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε αυτό το πέμπτο κομμάτι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Μόνο το binding, binding, το binding Παράγραφος 6 με κατατμήματα ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ και η Φιλελεύθερη. Υπέρ της παραγράφου 6 στην αρχική της μορφή, κατά, αποχές, απορρίπτεται. άρα δεν εγκρίνεται η αρχική μορφή του έξι. Τροπολογία 7 μπουλόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 λάμπερτ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8 τροπολογία 9 μπουλόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Yes, amendment 1 has been withdrawn. Ναι, η ένα αποσύρθηκε. Η τροπολογία ένα αποσύρθηκε. Alors, Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 30 υπέρ 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήριο στον εισηγητή μας. Συγγήτρια, εισηγήτρια, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, Συγγήτρια. Νομίζω ήταν και η πρώτη έκθεσή τη ε, στην Επιτροπή μας. Πάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της επιστολής ε, προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη δεύτερη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίπτωση της Δανίας. Υπέρ Νομίζω ότι καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Προπολογισμών στις 12 Ιουλίου. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση κινητοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται εδώ για μία περίπτωση ε, ισπανική στην Αραγωνία, στον τομέα των, ε, της κοδόμησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 30 υπέρ, μία ψήφος κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται η επιστολή. Θα θυμάστε ότι είχαμε ψηφίσει τις ε, τροπολογίες της κυρίας ε, ε, της, της έκθεσης κυρίας Σταϊνού, αλλά δεν είχαμε ψηφίσει το νομοθετικό ψήφισμα. Δεν το είχαμε ψηφίσει και επομένως πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικός το νομοθετικό ψήφισμα που έχει να κάνει με την έκθεση της κυρίας Στάινρουκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Το νομοθετικό ψήφισμα εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Στάινρουκ. Η έκθεση Χάντελ τώρα. Είστε όλοι έτοιμοι να την εξετάσουμε? Θα ήθελα να ζητήσω από την ομάδα Γκουέ, κυρία Τσούμπερ, ποιος θα αντικαταστήσει τον κύριο Χάντελ. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να διακόψουμε. Που δεν είναι ποτέ ευχάριστο, ούτε για μας, ούτε για τους διερμηνείς. Και για κανέναν από το προσωπικό που μας συνοδεύει. Υπάρχει κάποιος από την Γκουέ. Η κυρία Τσούμπερ έρχεται, μου λένε, οπότε προτείνω να την περιμένουμε λίγο. Euh, Διακόπτουμε λιγάκι μέχρι να έρθει η κυρία Τσούμπερ.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. για να επαναλάβουμε τις εργασίες μας και να περάσουμε στην εξέταση του σημείου 20 της ημερήσιας διάταξης όπως το είχαμε αποφασίσει, που αφορά την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης του κυρίου Τόμας Χέντελ προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ σε σχέση με την πρόταση οδηγίας ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για, την, για τις συμβάσεις παραχώρησης. Η κυρία Τσούμπερ αντικαθιστά τον κύριο Χέντελ γιατί ασθενεί. Κυρία Τσούμπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για λόγους υγείας, ο συνάδελφος Χέντελ δεν μπορεί να είναι σήμερα παρόν, οπότε θα κάνω εγώ αυτή την παρουσίαση που είχε ετοιμάσει ο ίδιος. Ο συνάδελφος προτείνει την απόρριψη της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και στην γνωμοδότησή του αναφέρει μία σειρά επιχειρημάτων ε, που θα παριθμίσω και εγώ αμέσως. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είναι μείζον για τον εισηγητή είναι το εξής. Αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις στις δημόσιες διοικήσει, με αυτή την πρόταση για τι συμβάσει παραχώρηση θα βρεθούν σε μια κατάσταση όπου πολύ συχνά θα υποχρεούνται να επιβάλλουν την ιδιωτικοποίηση πολλών υπηρεσιών κοινή ωφελία. Μάλιστα αυτή η πρόταση οδηγίας αναφέρει ότι το σχετικό κριτήριο που θα ακολουθείτε είναι η πλέον ωφέλιμη οικονομική πρόταση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στις δημόσιες διοικήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, μπροστά σε μια διαδικασία υποχρεωτικής ανάθεσης, να βρεθούμε όλο στην κατάσταση αυτή, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ανάθεση. Θα πρέπει λοιπόν οι δημόσιες υπηρεσίες ή να προβαίνουν σε προτάσεις ε, που να δίνουν πιο οικονομικό κέρδος από ότι οι ιδιωτικές εταιρείες και ε, με αυτόν τον τρόπο να υπονομεύουν σε ένα βαθμό το κοινωνικό κράτος. Ο συνάδελφός μου λοιπόν λέει ότι σε θέματα παραχωρήσεων με τέτοιου είδου ρυθμίσεις δεν πρόκειται να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά δεν είναι αυτός ο τρόπος για την εξυγίανση της οικονομίας. Με άλλα μέτρα εξυγίανσης και όχι με τέτοια συμπίεση των δημόσιων οικονομικών στοιχείων. Από την άλλη, γνώμη του συναδέλφου μου είναι ότι αυτή η πρόταση δεν δίνει καμία ασφάλεια δικαίου. Καθώς έχουμε και πολλές αναφορές που αποκλίνουν από την νομολογία του ΔΕΚ και μάλιστα το κριτήριο μεταφοράς του κινδύνου κατά τον αδελφό μου είναι ανεπαρκή. Δηλαδή, σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας κάποιου αναδόχου, τι θα συμβεί. Πολύ συχνά σε τέτοιε περιπτώσεις, το κράτος θα πρέπει να ε, μπει πάλι στο σκηνικό για να εγγυηθεί τον κίνδυνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή, αφαιρεγγιότητας, ε, των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν λάβει την ανάθεση. Θεωρούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών δεν εξασφαλίζονται. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την Επιτροπή μας, θέλω να αναφέρω εδώ. Αναφέρομαι στην δυνατότητα ε, υπαναχώρησης ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων ιδίως ό,τι αφορά την μείωση των μισθών, στην ε, ενίσχυση των περιπτώσεων κοινωνικού και εργασιακού dumping, κάτι που είναι βεβαίως εις βάρος των εργαζομένων, και όλα αυτά για να ασκηθούν πιέσεις στις τιμές, ώστε να μεσο μειοδοτικών διαδικασιών να γίνονται αυτές οι παραχωρήσεις. Όλα αυτά, αυτές οι διαδικασίες, είναι εις βάρος πάντων των εργαζομένων. Εργαζόμενοι είτε των εταιριών αναδόχων, είτε των δημοσίων υπαλλήλων, αυτών των δημοσίων υπηρεσιών που θα εκχωρούνται στον ε, ιδιωτικό τομέα. Οι δημόσιες υπηρεσίες, θεωρεί ο θα πρέπει να παρέχουν κοινά συλλογικά αγαθά προς τους πολίτες και να μην υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες του ανταγωνισμού που διέπουν γενικά την αγορά. Για αυτούς τους λόγους, για αυτά τα επιχειρήματα και άλλα που απαριθμούνται επίσης σε αυτή τη γνωμοδότηση του κύριου Χέντελ, προτείνω την απόρριψη της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμβάσεις παραχώρησης. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Λίζια Ρόν και θα κάνω μια δήλωση για λογαριασμό της. Τη διαβάζω. Έχει τίτλο «Γενικά σχόλια» στα αγγλικά. Να πω καταρχή η πρόταση 6.2 επιτέλους δημιουργεί κοινό πλαίσιο για τις αναθέσεις. Κάποιες παραχωρήσεις μπορεί να επηρεάζουν την αγορά. Γι' αυτό πρέπει να υπογραμμίζουμε τις ανάγκες σαφών κοινών κανόνων όλων των εμπλεκομένων, ενθαρρύνοντας ενιαία προσέγγιση στα 27 κράτη-μέλη. Δεύτερο σημείο, βελτίωση της διάκρισης μεταξύ παραχωρήσεων και συμβάσεων υπηρεσιών. Οι περισσό, τα περισσότερες συμβάσεις έργου συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις υπηρεσιών και είναι δύσκολο γι' αυτό να διακρίνουμε ποια κατηγορία εμπίπτει σε, ποια σύμβαση. Τρίτον, διευκρίνηση, διευκρίνηση της ε, διάρκειας ε, όπως προβλέπεται από την πρόταση που λαμβάνει υπόψη μόνο τη φάση διαχείρισης του έργου και οι υπηρεσιών και όχι τη φάση της δημιουργίας της δραστηριότητας. Τέταρτον, σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την ελευθερία επιλογής αν θα ε, κάνουν μόνες τους ε, τη δουλειά και τις υπηρεσίες ή αν θα παραχωρήσουν σε τρίτους. Αν αποφασίσουν να εμπιστευτούν την υλοποίηση σε τρίτους, θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ορίζουν τα νομικά μέσα που θα, που θα ισχύουν άδεια, δημόσια σύμβαση ή παραχώρηση. Σημείο 5. Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Ε, ενθάρρυνση της αυτοπιστοποίησης επειδή ως επιτοπλίστων συνεπάγεται σημαντικά ωφέλη και για τις κατασκευαστικές αρχές και για τους αναδόχους και για τους, ε, τις οικονομικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. κυρία Στρέλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δικαιολογήσω το γεγονός ε, ότι ήμουν απούσα στην αρχή της συζήτησης. Αλλά τώρα έλαβα γνώση της αλλαγής ε, ε, στην ημερήσια διαταξή. Αυτό το σημείο προβλέπεται να συζητηθεί το απόγευμα. Έπρεπε να είμαι παρούσα στις ψηφοφορίες ε, στην Επιτροπή Γυναικών και Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τούτου λεχθέντος, σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση και ως σκιώδης ηγήτρια της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς στηρίζουν σε ένα βαθμό την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές ρυθμίσεις για αυτές τις παραχωρήσεις και υπάρχει ένας βαθμός αδιαφάνειας στις δικασίες παραχώρησης. Αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην γενικότερη αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας αυτών των δικασιών. Μάλιστα υπάρχουν α, μελέτες σε συγκεκριμένους επιμέρους τομείς που μιλούν για ένα συνολικό όγκο 188 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις παραχωρήσεις ανάμεσα στο 2009 και το 2011. Επίσης, θέλουμε να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να απολαμβάνουν υπηρεσίες ποιότητας στις καλύτερες δυνατές τιμές, χωρίς αυτό να προκαλεί ε, στρεβλώσεις ε, στην εσωτερική αγορά. Υπ' αυτή την έννοια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να μπορεί να διασφαλίσει την σύγκληση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα βεβαίως να αγκιάται την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κυκλοφορία μάλλον αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 27. Επίσης, αυτή η οδηγία θα πρέπει να ε, προστατεύσει ε, την απασχόληση ποιότητας και να συμβάλλει στην πάταξη του κοινωνικού ντάπινγκ, ειδικά στις συνολογικέ περιπτώσεις. Τα κοινωνικά κριτήρια ε, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη σε αυτές τις διαδικασίες ε, παραχώρησης. Ε. Επίσης, να πω εν τέλει ότι θεωρούμε το εξή. Δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομικά, οικονομολογικά, αν θέλετε, τα κριτήρια αλλά και άλλοι παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία, παράγοντες όπως ήδη ανέφερα, αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια της βιωσιμότητας, ε, της ποιότητας και προσπελασιμότητας των υπηρεσιών προς τον χρήστη. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πολύ σημαντικό τομέα πολιτικής στον οποίο θα πρέπει να δοθεί προσήκουσα προσοχή καθώς μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών προσφέροντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Συμφωνείτε λοιπόν με όλους όσους πήραν το λόγο αυτό το, σε αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Τσούμπερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω μόνο θα ήθελα τους ε, ομιλητές. Κατέγραψα τα σχόλια και θα τα διαβιβάσω στον συνάδελφο τον κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Προτείνω τότε μέχρι τις 17 Ιουλίου κατάθεση τροπολογιών, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε 18 Σεπτεμβρίου. Συμβιβαστικές 8 Οκτωβρίου, να ψηφίσουμε 9 Οκτωβρίου. να έχουμε λίγο χρόνο ανάμεσα στις συμβιβαστικές ε, και στην ε, ψηφοφορία, γιατί 10 ή 13 Δεκεμβρίου ψηφίζει η ΙΜΚΟ. Οπότε εμεί θα είμαστε πολύ μπροστά στη συζήτηση. Λοιπόν, μπορούμε να διακόψουμε την συνεδρίασή μας για ένα τέταρτο. Αλλού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, όπως είχαμε πει, ο κύριος Φιλίπ ε, Ντεμπούκ δεν χρειάζεται να σας τον παρουσιάσει κανείς. Ε, είναι ο Γενικός Διευθυντής ε, της Business Europe εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Θέλησε λοιπόν να ε, μας μιλήσει σήμερα για να μας πει την άποψη ε, των εργοδοτών σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Είχαμε πολύ συχνά ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και συμμετείχαμε στην επεξεργασία ενός ψηφίσματος ε, για το ε, θέμα αυτό εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του ΕΑΡΙΝΟΥ. Βέβαια, δυστυχώς Υπήρχαν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα να συζητηθούν σε αυτό το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά η απασχόληση παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εξού και η σημασία της ε, δικής σας άποψης, ε, την οποία θα μοιραστείτε μαζί μας, ε, της άποψής σας ως σημαντικής οργάνωσης. Κύριε Ντεμπούκ, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να ε, πάρω το λόγο σήμερα στην Επιτροπή σας. Είναι μεγάλη η επιθυμία μου να πάρω το λόγο εδώ. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχετε συζητήσει πολύ, πολλές φορές το θέμα της, ε, του πακέτου για την απασχόληση και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να, να παρουσιάσω και τις απόψεις της Business Europe που γνωρίζετε ότι εκπροσωπεί όλους ε, τους, ε, όλες τις οργανώσεις εργοδοτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, θελήσατε να με παρουσιάσετε, διότι πολλά χρόνια είμαι διευθυντής της Business, ε, ε, της business Europe, όμως για μερικούς μήνες ακόμη, γιατί όπως ανακοίνωσα θα αποχωρήσω στο τέλος της χρονιάς, μετά από μια πολύ ενθουσιώδη και μακρόχρονη καριέρα στην Business Europe. Θα ήθελα λοιπόν να επωφεληθώ και να ευχαριστήσω και την δική σας Επιτροπή για όλες τις συζητήσεις και επαφές που είχα και με εσά ως πρόεδρο Πρόεδρο αλλά και με ε, πολλά από τα μέλη της Επιτροπής σας. Τώρα θα θέλω να περάσω στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω σας προσωπικά και την Επιτροπή σας για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Πριν την τελευταία σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είχε ως αντικείμενο την εξέβρεση λύσεων για την Ευρωζώνη, το νόμισμα του ευρώ και να καταλήξει κάποιες στιγμές συνθήκες για μία πολιτική στρατηγική ανάπτυξης. Πριν λοιπόν από αυτό, εμείς ε, εκπονήσαμε ένα σύντομο φυλάδιο προσβάσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά και στο website μας με τίτλο «Πώς μπορεί κανείς να αναπτυχθεί και να οδηγηθεί σε μεγέθυνση και να βγει έξω από την κρίση». Ε, δεν θέλω να μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες, γιατί τα πιο πολλά και τα αναφέρουμε σε αυτό το φυλάδιο. Πιστεύουμε εδώ και χρόνια ότι μόνο με μία στρατηγική ανάπτυξης και με μία γέφυνση της οικονομίας μπορούμε να επιτύχουμε τα πεδιοκόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ήδη έχουμε πει ότι για να επιτύχουμε τους στόχους στρατηγικής 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να μπορέσουμε με βιώσιμο τρόπο να διαφυλάξουμε τα κοινωνικά μοντέλα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη μας, χρειάζομαστε κατά μέσο όρο μία ανάπτυξη 2,5% ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μπορούμε να ε, επιτύχουμε την πλήρη απασχόληση του 2020. Βεβαίω η ανάπτυξη είναι ένα στοιχείο, ένα παράγοντα. Μπορούμε επίση να συζητήσουμε και τα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά πέρα από την ανάπτυξη, ή μάλλον για να επιτύχουμε τους στόχους της ανάπτυξης, θα πρέπει να πληρούμε και κάποιους άλλους όρους που θα αναφέρω σε λίγο. Σε ό,τι αφορά το πακέτο για την απασχόληση, είναι προφανές ε, ότι χρειάζεται μια ανοιχτή συζήτηση πρώτα απ' όλα με τον Επίτροπο Άντορ, ο οποίος είναι αρμόδιος με τα θέματα κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης, όπως και με τους συναδέλφους κοινωνικούς εταίρους, ε, με τους οποίους είχαμε μακρές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω ότι για να έχουμε ανάπτυξη και δημιουργία τη εργασίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να σκέψουμε πάνω στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα θα δημιουργήσει τι συνθήκε για αύξηση των θέσεων εργασία, για ανάπτυξη και θα αποτελέσει το μοχλό για την χρηματοοικονομική και δημοσιονομική ε, βελτίωση κατάστασης ε, στα κράτη-μέλη. Το κόστος της εργασίας βεβαίως είναι ένα στοιχείο κλειδί και σίγουρα είναι μία καλή προσέγγιση για να δούμε το θέμα σφαιρικά. Αυτό ήδη γίνεται σε πολλά Το κόστος της εργασίας δεν είναι αναγκαστικά το μισθολογικό κόστος, καθώς το κόστος εργασίας μπορεί να μειωθεί μειώνοντας τις εισφορές των εργοδοτών ώστε να αποδοθούν κίνητρα στην εργοδότηση, την ε, προσλήψεις, καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τη Για τη δημιουργία της εργασίας η Κομισιόν προτείνει τρεις ε, τομείς όπου μπορούμε να ε, δουλέψουμε περαιτέρω. Τρεις μίζονες τομείς αλλά διέπονται από διαφορετικά οικονομικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα η υγεία Δεύτερον, η πράσινη οικονομία, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και ο τρίτος τομέας είναι η κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας, το ICT. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το ICT. Αυτός ο τομέας είναι ένας ευρύτατος τομέας δραστηριοτήτων που υπάρχει και μέσα στα πλαίσια και των άλλων τομέων. Είτε μιλάμε για τον δημόσιο, είτε για τον ιδιωτικό τομέα καθώς ένα μεγάλο κομμάτι και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ε, διέπονται από τις εξέλιξεις στην πληροφορική τεχνολογία. Και το ψηφιακό θεματολόγιο προκειμένου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί ανοίγει νέε λεωφόρους που συνδέονται με το διαδίκτυο και σχετικές δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι εδώ θα σημαντικά σε σχέση με τις ΙΠΑ για παράδειγμα. Και όταν μιλώ για... το μάλλον ότι υπολοιπόμεθα, μιλάμε για ένα μεγάλο κενό. Ιδίω αν δείτε τα θέματα της ψηφιακής κοινωνίας. Θα δείτε ότι οι πιο πολλές εξελίξεις, τα πιο πολλά επιτεύγματα λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όμως, το ICT από τη μία κινητοποιείται από τις ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή δεν χρειάζονται δημόσια κονδύλια. Είναι οι δυνάμεις της αγοράς που θα λειτουργήσουν, αρκεί βεβαίως να υπάρχει ένα ορθό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την ε, πράσινη οικονομία, πράγματι, Χρειάζεται να απελευθερώσουμε την οικονομία μας από τη χρήση του άνθρακα. Ε, εμείς στην Business Group το, το επιδιώκουμε αυτό. Πάντοτε στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου της ανταγωνιστικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Τα θέματα του κλίματος είναι εξορισμού θέματα παγκόσμια. Και εδώ υπάρχουν λεωφόροι που σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχει το πρόγραμμα ETS, υπάρχουν οι στόχοι του 2020 για την μείωση των εκπομπών λοιπόν, του άνθρακα και για να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους, θέλω να πω την οπτική γωνία ε, της βιομηχανίας, κατά πάσα πιθανότητα θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι του 2020. Όμως επήγει, αυτό το θέμα, κάτι που είπαμε και πρόσφατα στην Κομισιόν. Επήγει λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε μετά το 2020 ποιοι θα είναι οι στόχοι μετά και ποιε θα είναι οι πολιτικές μετά το 2020, διότι για του κύριους παίκτε, ιδίω για τις βιομηχανίε εντάσεις ενέργειας, το 2020 είναι ήδη αύριο. Η βιομηχανία επενδύει με ορίζοντα δεκαετίας, εικοσαετίας και πάνω. Οπότε εξορισμού αυτή τη στιγμή κοιτούν πέρα από το 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, υγεία και την ε, κοινωνική περίθαλψη, εδώ ε, θα πρέπει να κάνουμε μία εισβάθος ζήτηση. Ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη. Μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε συμπράξεις δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Πώς θα αναπτυχθεί αυτός ο τομέας που για πολλούς λόγους, είτε μιλάμε λόγω τεχνολογικών εξελίσσεων, αλλά και σε επίπεδο ζήτηση και σε επίπεδο προσφοράς και λόγω των δημογραφικών εξελίσεων έχουμε να κάνουμε ένα τεράστιο πεδίο ε, το οποίο θα πρέπει να οργανώσουμε, να οργανώσουμε καλά. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τους άλλους τομείς, αλλά δεν θέλω να τους αναπτύξω όλους. Εγώ εστιάζω στους τρεις τομείς ε, που προτάσει η Κομισιόν. Πάντως υπάρχει ένα κύριο ζήτημα για το οποίο θέλω να τοποθετηθώ εδώ νόπιόν σας. Αν ρωτήσουμε τα μέλη μας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις ε, που βρίσκονται μπροστά μας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο. Ναι, αμέσως σκεφτόμαστε τον χρηματοοικονομικό τομέα, τον ανταγωνισμό με την Κίνα, τα θέματα απορρίθμισης κτλ. Αλλά μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, ποια είναι η κύρια πρόκληση που πιστεύετε ότι έχετε να αντιμετωπίσετε τότε η απάντηση είναι η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Εργατικού δυναμικού υψηλή ειδίκευση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε μια ευρία γκάμα επαγγελμάτων ώστε να δούμε πού υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στην ε, προσφορά και στη ζήτηση θα πρέπει να δούμε εν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα θέματα μαθητείας. Στις χώρες εκείνες που υπάρχουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, με αποτελεσματικό τρόπο, βλέπουμε να μειώνουν τα ποσοστά ανεργίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τους επιμέρους τομείς και τις συνέπειες, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Και στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί με τα συνδικάτα ήδη από το 2007, πριν δηλαδή την κρίση, και εξετάσαμε πώς θα λειτουργούν οι αγορές εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. και καταλήξαμε σε κάποιες αξιολογήσεις, αποτιμήσεις ε, της κατάστασης και προβήκαμε και σε κάποιες συστάσεις. Βεβαίως εδώ υπάρχουν και ε, αφιστάμενες απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσει. αλλά τελικά καταλήξαμε ε, από κοινού στον όρο flexicurity, ε, ευελιξία και ασφάλεια στην εργασία. Και θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να προαχθεί στα κράτη-μέλη. Βεβαίω, για να μην υπάρχουν παρανοήσει, όταν μιλούμε για ευελιξία και ασφάλεια στην εργασία, flexicurity, και βεβαίω ξέρουμε ότι τα συνδικάτα δίνουν πιο πολύ έμφαση στην ευελιξία και όχι στην ασφάλεια, και θεωρούμε ότι αυτό είναι λανθασμένο. Εμεί θέλουμε ευελιξία για τι επιχειρήσει, αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια για του εργαζομένου. Όμως η ασφάλεια σε ένα κομμάτι βεβαίως είναι η οικονομική εξασφάλιση όταν χάνουν μια θέση εργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ασφάλεια. Αυτό που καλούμε, αποκαλούμε ως απασχολησιμότητα. Τι σημαίνει όταν χάνεις με τις εργασίες να μπορείς πιο εύκολα να βρίσκεις μια καινούρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ασφάλειας. Για να κινητοποιηθεί η έργα εργασίας. τι σημαίνει ουσιαστικά τι θέλουμε να επιτύχουμε όταν κανείς χάνει μία θέση εργασίας να μπορεί να βρίσκει μία άλλη, διότι η οικονομία έχει μία δυναμική, είναι ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται συνεχώς ανα, αναδιαρθρώσεις, συνεχώς αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεν ευελιξία, ασφάλεια δε. Και αν θέλετε να αντιστρέψω και τις έννοιες. Κάτι γνώμη μας, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και ασφάλεια για τους εργαζόμενους τους. Στην οικονομία της γνώσης, ξέρετε, μπορεί πριν από 20 χρόνια να ίσχυε, δεν ίσχυε όμως σήμερα, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να αντικατασταθούν μια ανοιχτή. Οι εργαζόμενοι είναι δεσμευμένοι, αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους ε, και σε μια οικονομία υπηρεσιών είναι απαραίτητη η ασφάλεια και για τους εργαζόμενους. Η έννοια τη ευελιξία επίση δεν είναι πολύ σαρνητική. Πολύ συχνά και οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία. Λοιπόν, οι εθνικέ μεταρρυθμίσει είναι κλειδί ε, στην λύση των προβλημάτων, α, περισσότερο σήμερα από ποτέ, στην παρούσα οικονομική συγκυρία και για να ανακοφιστούν ε, χώρε που αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη οικονομική πίεση. Πρόσφατα έχουν γίνει πολλά, αλλά και νωρίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία, αλλά και πιο πρόσφατα σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και αλλού. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένας κινητήριος μοχλός για τον εξυγχρονισμό της οικονομίας και της αγοράς εργασίας με ισόρροπο τρόπο. Υπήρξαν και υπάρχουν ε, κάποιες προτάσει στο τραπέζι για τις ε, συμβάσει απασχόλησης και τι είδου ε, συμβάσει απασχόλησης θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να προωθήσουμε. Θέλω πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Eurofound, το Ίδρυμα του Βουβλίνου δηλαδή, σχεδόν το 85% των συμβάσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι παραδοσιακές κλασικές συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες ε, μορφές ε, συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας. Και θέλουμε να κρατήσουμε και αυτές τις άλλες μορφές εργασίας. Αυτό είναι στοιχείο ευελιξίας, αλλά ταυτόχρονα και ένας τρόπος εξέβρεση εργασίας για πολλούς ανθρώπους και ένας τρόπος ε, διείσδυσης στην αγορά εργασίας για πολλούς. Άρα δεν μπορούμε συνεχώς ε, να στιγματίζουμε τέτοιες μορφές απασχόλησης λέγοντας ότι αυτές είναι οι επισφαλείς θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη επισφάλεια είναι η ανεργία. Οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ώστε να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας είναι κάτι που πρέπει να χαιρετήσουμε. Ήδη είπα κάτι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το μέλλον αλλά και για το παρόν. Αυτό που αναφέρεται και στον γράφο της Κομισιόν ως αναντιστοιχεία δεξιοτήτων και αναγκών. Ήδη έχουμε εκατάδες χιλιάδες κενές εργασίες ακριβώς γιατί υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην ζήτηση και τις δεξιότητες και αυτό δεν αφορά μόνο τις πλέον εξειδικευμένες θέσεις αλλά και σε όλη την γάμα, σε όλη την κλίμακα α, απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο με την εκπαίδευση την, και την κατάρτιση. Στην Business Europe έχουμε κάνει σημαντική δουλειά πρόσφατα στο θέμα των ε, δικών συστημάτων ε, εκπαίδευσης, κατάρτισης ε, με προγράμματα μαθητείας. Θεωρούμε ότι αυτά τα δικά συστήματα πρέπει να εφαρμοστούν παντού. Θεωρούμε ότι τα κράτη εκείνα που αποτελεσματικά εφαρμόζουν τέτοια συστήματα διοικής ε, μάθηση και κατάρτιση αναφέρομαι σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτέ λοιπόν οι χώρες έχουν εργαζόμενου καλύτερα εκπαιδευμένου, καλύτερα καταρτισμένου και μικρότερο ποστό ανεργίας μεταξύ των νέων. Διότι ειδικά σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της ανεργίας των νέων, είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να εκριζώσουμε πλήρω, διότι όταν ο, ο μέσο ευρωπαϊκό όρο ανεργία μεταξύ είναι 25%, αυτό τι σημαίνει, ότι θυσιάζεται μια γενιά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στις χώρες εκείνες όπου ε, προβλέπονται προγράμματα μαθητείας ε, και ειδικών συστημάτων κατάρτισης, ο μέσος όρος ανεργίας είναι πολύ χαμηλότερος. Η ανεργία των νέων, όπως δείχνουν οι στατιστικές, είναι ας πούμε στα 16 με 18 και 25. Συνδέεται και με την εκπαίδευση εκείνη την εποχή. Στη Γερμανία είναι 4%, ενώ είναι 25% στην Ισπανία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κέριο ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Για ε, διακυβέρνηση, ναι, οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να ενταχθούν στη νέα διακυβέρνηση, την ενωσιακή διακυβέρνηση. Δεν σημαίνουμε τι σημαίνει αυτή η νέα ενωσιακή διακυβέρνηση. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά έχουμε ε, συμφωνήσει με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες, τους εργοδοτικούς φορείς, να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες αυτό το θέμα μετά το καλοκαίρι αμέσω για να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ή δυνατόν κοινέ προτάσεις. Ξέρετε ότι ήδη συμμετέχουμε στο, στην τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής δύο φορές το χρόνο πριν από την αερινή σύνοδο και πριν από την ε, σύνοδο του Οκτωβρίου Έχουμε και αυτό που λέμε μακροοικονομικό διάλογο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο όπου συζητούμε θέματα οικονομικά και νομισματικά και τις πολιτικές μας και τον αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο και αν μπορεί ο αντίκτυπος να βελτιωθεί. Όλα αυτά θα τα δούμε πολύ θετικά. Αυτό που είναι σημαντικό για μας τουλάχιστον είναι ότι η ενωσιακή διακυβέρνηση θα ενισχυθεί. Θα πρέπει να συζητήσουμε όλα τα δομικά στοιχεία των συμπερασμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι βεβαίως πολύ σημαντικά. Αυτά είναι κάποια γενικότερα σχόλια. Τώρα, εις ό,τι αφορά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, εγκρίνατε στην Επιτροπή αυτή. Όπως σας είπα, εγκρίνουμε και χαιρετίζουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μειωθεί ο φόρος επί της εργασίας με τρόπο που να μην επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Για τη συμβάσεις εργασίας χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αναγνωρίζει το Κοινοβούλιο ε, την ανάγκη να στηρίξουμε την, ε, με νομοθετικά μέτρα για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τα προγράμματα θέσεων εργασίας είμαστε πολύ κοντά γιατί συμφωνούμε και εγώ και εμείς με το Κοινοβούλιο που λυπάται διότι δεν υπευλήθησαν από πολλές χώρες εθνικά σχέδια θέσεων εργασίας ως μέρος του προγράμματος του 2012 και αυτό είναι κρίμα γιατί όσο πιο σαφώς θα περιγραφεί σε εθνικό επίπεδο η κατάσταση τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα δείξουν και οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που θα προσλαμβάνουν τότε κόσμο αφού θα ξέρουν σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν. Τώρα για τον ελάχιστο μισθό, το βασικό μισθό το αφήνουμε στα κράτη-μέλη για να το χειριστούν. Αυτό είναι ένα ε, στοιχείο το οποίο είναι τόσο εδρεωμένο στο εθνικό σύστημα που δεν είναι κάτι που μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνούμε για την επιχειρηματικότητα με τις απόψεις σας. Βεβαίως πρέπει να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα όχι μόνο για τους νέους, αλλά για ανθρώπους αργότερα στη σταδιοδρομία τους, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσουν μια επιχείρηση, για την πρακτική εξάσκηση και εκεί πρέπει να κάνουμε κάποια δουλειά και να αφιερώσουμε κάποια κονδύλια για να τη χρηματοδοτήσουμε. Συμπερασματικά λοιπόν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε περισσότερα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κρίστενσεν και μετά Κορνέλισεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιλίπ Ντεμπούκ για την παρουσίαση του πακέτου απασχόλησης και την άποψη του Business Europe. Συμφωνώ με όλα σχεδόν αυτά που είπατε για την αναπτυξιακή στρατηγική και το πακέτο απασχόλησης, ώστε να ε, υλοποιήσουμε τη στρατηγική 2020. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, σε όλη την Ευρώπη όμως, υπάρχουν φόβοι. Πάντα υπήρχε συνεργασία ούτως ώστε στην αγορά εργασίας να υπάρχει ένα επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες τους και ένα κοινωνικό μοντέλο για το οποίο μπορεί να είμαστε περήφανοι. Τα μέτρα λιτότητας απείλησαν το κοινωνικό μοντέλο και το έθεσαν ενώπιον τεραστίων πιέσεων. Αν δούμε την κατάσταση σήμερα, γνωρίζουμε ότι σχεδόν παντού στην Ευρώπη όλη η αύξηση της απασχόλησης ε, περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ορισμένου χρόνου και είναι χειρότερες οι συνθήκες εργασίας σε σχέση με αυτούς που έχουν συμβάσει ορίστου χρόνου. Είπατε ότι ένα πρόβλημα είναι το κόστος εργασίας, το εργασιακό κόστος και είπατε ότι δεν είναι αναγκαστικά η συνιστόσα των μισθών, αλλά και οι κοινωνικές εισφορές από τις εταιρείες των εργοδοτών κλπ. Το σκέφτηκα αυτό το θέμα. Ίσως ε, ένα από τα προβλήματα στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε διαφορετικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία. Στις ε, σκανδιναβικές χώρες ε, πληρώνουμε από τους φόρους την κοινωνική πρόνοια. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης πληρώνουν οι εταιρείε μέσω των κοινωνικών εισφορών. Όταν μιλάμε για τη δημιουργία περισσότερης εκπαίδευσης για τους νέους, ε, καλύτερης εκπαίδευσης κατάρτισης του εργατικού δυναμικού μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, τότε δυσκολεύονται τα πράγματα, γιατί τότε θα σκεφτεί ο καθένας «Α, θα επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο κόστος οι επιχειρήσεις σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ σε άλλες θα πληρώνονται όλα αυτά μέσα από τους φόρους». Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Μιλήσατε και για την ευελιξία με ασφάλεια. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στη σωστή ισορροπία σήμερα. Σε πολλές χώρες οι άνθρωποι χρειάζεται να δουλεύουν δύο δουλειές για να φροντίσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Ε, δουλεύουν ως φτωχοί και δεν είναι αυτό που θέλουμε, σίγουρα αυτό στην Ευρώπη, θέλουμε μισθούς και ημερομίσθια για να συντηρούμεθα και να προσφέρουμε και κάτι στις οικογένειές μας. Μιλήσατε για το διοικό σύστημα εκπαίδευσης και συμφωνώ ότι είναι πολύ καλό σύστημα γιατί υπάρχει θεωρητική εκπαίδευση στις σχολές και η πρακτική εκμάθηση στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εκπαίδευσης ιδιαίτερα των νέων. Και αν δούμε τους νέους, αυτοί βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο σήμερα, διότι δυσκολεύονται να βρουν θέση απασχόλησης. Τι προτάσεις έχετε, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε περισσότεροι ε, νέοι άνθρωποι να μπουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Κορνέλισεν και μετά Ρή. Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την παρέμβασή σας. Αισθάνομαι όμως ότι έλειπαν ε, κάποια ζητήματα. Τρία ζητήματα θέλω να θέσω. Πρώτον, είπατε ότι η μεγαλύτερη επισφάλεια στην εργασία είναι η ανεργία. Εγώ διαφωνώ η, η φτώχεια, η ένδια μέσα στην επασχόληση είναι η μεγαλύτερη επισφάλεια. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν 80 ώρες την εβδομάδα ε, και δεν ε, ξεπερνούν καν το όριο της φτώχειας. Διότι αυτό δεν δίνει καν μία διέξοδο την ελπίδα ότι αν δουλέψω σκληρότερα θα βγω από τη φτώχεια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα αυτό τις φτώχειας ε, στην εργασία είναι κάτι που θα πρέπει να ε, δείτε. Ε, Μιλήσατε για την αντιστοιχία στις, στην κατάρτιση στις δεξιότητες. Κοιτάξτε, σε μία κοινωνία σε εγκύρανση αυτό το πρόβλημα θα οξύνεται όλο και περισσότερο. Η κινητικότητα στην εκπαίδευση για κατάρτιση είναι σημαντική. Αυτό που μου λείψε από τοποθέτηση σχετικά είναι η θέση και ο ρόλος των εργοδοτών αντιμετώπιση των στερεοτύπων ε, διακριτικής μεταχείρισης, διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικία συχνά, καθώς οι επιχειρηματίες δεν ε, προσλαμβάνουν Ρωμά, μετανάστες, άτομα αναπηρίες, γυναίκες κτλ. Πολλοί συνεχίζουν να προτιμούν το πρότυπο ε, του λευκού άνδρα 25-45 ετών. Ε, και επειδή αρχίζει να στερεύει αυτή η δεξαμενή, τι θα κάνουμε. ρωτιέμαι. το έχετε δει αυτό το θέμα. Τρίτο και τελευταίο, για τους μισθούς, κάτι που αναφέρεται και στις συστάσεις, όπως και στο πακέτο για την απασχόληση. Υπάρχει μεγαλύτερη συμμετρία στο τομέα αυτό, προς το παρελθόν. Δηλαδή, λέτε, ότι και οι γερμανικοί μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν. Αυτές, αυτά είναι οι συστάσεις. Εσείς μεταξύ ημών ε, εργοδοτών, επιχειρηματιών, πώς το βλέπετε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και τους μοχλούς προς τα πάνω. Ο κύριος Ωρή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή, κυρίως γιατί εμείς στο ΕΛΚ είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει ε, να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, γιατί είναι αρκετά χαμηλό το επίπεδο απασχόλησης στην Ευρώπη και πιστεύω ότι ο ιδιωτικός τομέας κυρίως μπορεί να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, ε, στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ότι πρέπει να ε, ενισχυθεί και η προσφορά. Βέβαια, αυτό σημαίνει εν μέρη συμμετοχή του κράτους. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πώς βλέπετε αυτήν τη διάκριση, αυτό το διαχωρισμό μεταξύ των ιδιωτικών επενδύσεων, των ιδιωτικών εταιριών ε, και του ρόλου του ε, κράτους που κατά τη γνώμη σας ε, θα ήταν ευπρόσδεκτος μάλιστα. Ειδικότερα όταν δεν καταφέραμε και πάρα πολύ καλά να βγούμε από την κρίση και μεγάλη συνέπεια αυτού είναι ότι είναι μεγάλη η δημοσιονομική πίεση, κάτι το οποίο παρεμποδίζει την οικονομική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των ε, εταιριών. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να εξεύρει λύσεις, όμως δεν είναι πολύ σαφές οι λύσει αυτές για μα Και να προσθέσω κάτι ακόμη, σε σχέση με τους τομείς ε, ε, στόχους που ε, εντόπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για, την ιδιωτική, για τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική πτυχή βεβαίως, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικές πτυχές επαρκώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης χρειάζονται βρεφονιπιακοί σταθμοί, χρειάζονται τέτοιου είδους λύσεις. Εσείς ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, για τον ε, ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι πρέπει βεβαίως να μειώσουμε το κάτι το οποίο ούτως ή άλλως στη δέσμη μέτρων ε, για την απασχόληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται. Αλλά ποιοι είναι οι τομείς ε, της οικονομίας ε, στους οποίους υπάρχει η αίσθηση του κατεπήγοντος και αναφέρομαι κυρίω στα κείμενα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αφορούν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι υπάρχουν περισσότερες πρωτοβουλίε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, μείωση του άχθου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο παρακολύει την ανάπτυξή τους. Βεβαίω, επί της αρχή, συμφωνούμε ότι ε, το βασικό μήνυμα είναι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτή την ανάπτυξη ε, σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες και την Κίνα. Μεγάλη πρόκληση για μας αυτό. Η κυρία Γιαζουβιέσκα. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορέσαμε να συναντηθούμε εδώ και να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Εσείς έχετε πολύ πείρα από τις συζητήσεις σας με τους ε, εργοδότες. Στο έγγραφο για τις μεταρρυθμίσεις η Κομισιόν συστήνει να υπάρχουν σε, στο σωστό επίπεδο οι μισθοί να διαμορφωθούν στο σωστό επίπεδο για την ανάπτυξη των εξαγωγών για την εσωτερική κατανάλωση. Είναι σημαντική συνιστόσα της πολιτικής ε, για την, ανάπτυξη. Συχνά όμως οι εργοδότες λένε ότι πρέπει να περικοπεί το κόστος εργασίας. Τώρα, αυτά τα δύο πώς μπορεί να συμβιβαστούν ως αντιτιθέμενες απόψεις και πώς να έχουμε σωστή αμοιβή για την εργασία, αλλά να βοηθήσουμε και τους εργοδότες να μειώσουν το εργατικό κόστος για να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή λοιπόν είναι η μία ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για ευελιξία στην αγορά εργασίας. Συχνά αυτό που καταλαβαίνουμε από την, ε, οι εργοδότες καταλαβαίνουν ότι η ευελιξία σημαίνει συμβάσεις εργασίας όχι πρότυπες. Οι νέοι μπορεί να πάρουν συμβάσεις εργασίας αλλά ε, είναι ανοιχτές και πολλές φορές μπορούν να, δεν μπορούν να ε, συμβιβάσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους εργοδότες ε, να ε, βελτιώσουν τις συμβάσεις που προσφέρουν. Επίσης ε, μιλάμε για την εκπαίδευση. Μ' αρέσει που και οι εργοδότες προσέχουν το θέμα αυτό της καλής εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι το βασικό αν θέλουμε να έχουμε ψηλά πρότυπα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για την αξιολόγηση από την πλευρά των εργοδοτών, των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση είναι καλοί, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Καμιά φορά ομολογώ ότι αμφιβάλλω. Συχνά χρησιμοποιούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να διεξαγάγουμε διάφορες καταρτήσεις. Αλλά οι ίδιοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι. Ούτε η κατάρτιση ε, στοχεύει στις ανάγκες των εργοδοτών. Και έχω ακόμα δύο ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Στο έγγραφο που ετοίμαζα όταν ε, εργαζόμουν ε, στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων αγοράς εργασίας, ε, ε, ε, προσφέρονται τράπεζες ορών εργασίας όπως θα εις λέμε. Υπάρχει αυτό στο σχέδιο της Κομισιόν. Αυτό το θέλουν οι εργοδότες, συμφωνούν. Τέλος, η Κομισιόν παρουσιάζει, αν δεν κάνω λάθος, έξι διαφορετικά ευρωπαϊκά οικονομικά μέσα ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτά τα ταμεία πώς τα αξιολογούν οι εργοδότες και τα χρησιμοποιούν καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τρεις ερωτησούλες. Το πρώτο θέμα το θέσατε ήδη. Πώς αξιολογείτε την ε, πρόοδο που πρέπει να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για, την, για τα στάζ, γιατί είναι κάτι ε, για το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υποβάλει πιο συγκεκριμένη πρόταση αν θέλουμε να συμφιλιώσουμε την ανάγκη στάζ για τους νέους για να τους δώσουμε τη δυνατότητα της μετάβασης από τον κόσμο της εκπαίδευσης ε, στον κόσμο της απασχόλησης, αν θέλουμε αυτό να το ε, συμφιλιώσουμε με τη μη χρήση ε, των στάζ για κοινωνικό ντάμπινγκ στην αγορά εργασίας, πρέπει να πλαισιώσουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα στάζ, αυτήν την εκμάθηση και πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες, ε, να ισχύουν οι ελάχιστοι όροι για τα κρατη γιατί το είπατε και εσείς, πρέπει να προβληματιστούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, τέλος πάντων πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα, δεύτερη ερώτηση. Θα θυμάστε ότι ο Μάριο Ντράγκη, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ήταν παροχημένο, είναι παροχημένο, ότι πρέπει κάτι άλλο να γίνει τέλος πάντων. Εσείς πώς ε, εκλάβατε αυτή την πρόταση, αυτή την ε, ε, τη θέση του κυρίου Ντράγκη, βρίσκω ότι ήταν λίγο άτοπο το να πει κάτι τέτοιο, μήπως είναι ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή ότι το, κοινωνικό, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι το κεφάλαιο το πιο πολύτιμο ε, των Ευρωπαίων ε, και όταν αναλογίζεται κανείς τις την θέση του Βρετανού οικονομολόγου που λέει ότι ε, οι κοινωνίες τις οποίες δεν υπάρχουν μεγάλες ε, ανισότητες είναι αυτές τις οποίες υπάρχει κοινωνικός διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος και το κοινωνικό μοντέλο είναι μια ε, ένας παράγων ισχύος και δεν είναι η στιγμή να το εγκαταλείψουμε. Τρίτη ερώτηση. Εδώ και στη Γαλλία που γνωρίζω καλύτερα υπάρχει μία έκκληση υπέρ της ε, ανάπτυξης. Ε, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το μοντέλο. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο βαθιάς αλλαγής ε, και ότι τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε δεν θα επιληθούν μόνο με την ανάπτυξη. Για δύο λόγους. Πρώτον, η περίοδος πριν από την κρίση δεν παρήγαγε τις απαραίτητες θέσεις ε, απασχόλησης, τις απαραίτητες για τις ανάγκες ευρωπαϊκής οικονομίας. Ξέρω ότι υπάρχει φθήνουσα δημογραφία κλπ. και ότι δεν θα έχουμε τόσο ανάγκη απασχόλησης. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Αυτό το επιχείρημα, α, αν έχουμε κάτω από 2% ανάπτυξη δεν έχουμε απασχόληση, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κανένας, ε, καμιά μηχανική σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ της ανάπτυξη και της απασχόλησης. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, αν δεν το ομολογήσουμε αυτό, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης στις δυτικές οικονομίες. Δεύτερο θέμα υπέρ αυτής της ανάπτυξη, δεύτερο επιχείρημα, ε, λέγεται ότι η νομισματική κατάσταση είναι εντελώ αντιπαραγωγική αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη. Υπάρχει μια τεράστια πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χαμηλά επιτόκια και λέμε ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση και κοινωνική. Μα όχι, αφού βλέπετε ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια και είναι και πολύ χαμηλά, χαμηλότερα από ποτέ τα ποσοστά ε, τη απασχόληση. Άρα λοιπόν αυτά τα χαμηλά επίπεδα ε, επιτοκίων ε, πρέπει κανονικά να, να, να κάνουν κάτι άλλο εκτό από το να δημιουργούν κερδοσκοπία. Θα πρέπει να δημιουργείται πραγματική οικονομία. Ξέρω ότι οι εργοδότες δεν τους αρέσει να μιλάμε για πραγματική οικονομία, αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα. Συμφωνείτε λοιπόν ότι το να λέει κανείς ότι είναι υπέρ τη ανάπτυξης, αν δεν υποστηρίζεται από μία ε, δυνατότητα προσανατολισμού, ε, ε, δεν μιλάω υποχρεωτικά για κίνηση κεφαλαίων, μία επίδραση τέλος πάντων στις στρατηγικές χρηματοδότησης ε, ε, ε, δεν θα ε, ανταποκριθούμε στι ανάγκες της οικονομίας και ε, στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το είπατε αυτό, δεν λέω, αλλά πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη, έτσι όπως τίθεται νομίζω ότι είναι μία παγίδα και ελπίζω να μπορέσουμε να την να, επεξεργαστούμε κάπως διαφορετικά την κατάσταση για να είναι πιο υποσχόμενοι στρατηγικές. Νομίζω ότι δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, οπότε να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Ένα τεταρτάκι έχετε στη διάθεσή σας. Ελπίζω ότι είναι επαρκή, επαρκές. Τι να σας πω, πολύ δύσκολο θα είναι να απαντήσω και στα δικά σας ερωτήματα μέσα σε ένα τέταρτο. Ναι, λέει η Πρόεδρος, ελπίζω πάλι να έχετε μια καλή ανάμνηση της ανταλλαγής απόψεων που κάναμε. Κοιτάξτε, ε, ελπίζω τα μέλη της Επιτροπής σας ε, να μου επιτρέψουν να απαντήσω πρώτα στο δεύτερο ερώτημα της Προέδρου σας, γιατί νομίζω ότι είναι κεφαλαιόδου σημασίας για το ε, υπόλοιπο της παρουσίασής μου και της επιχειρηματολογίας μου. Δεν θα αναφερθώ ε, σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στο διάλογο μακροοικονομικό που κάνουμε με τους κοινωνικούς εταίρους, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πολλά πράγματα λέγονται και είναι επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα, απαντώντας στο σχολείο να σας πω ότι στην Business Europe εμείς ε, υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το είπαμε, το ξανάπαμε, το γράψαμε, το ξαναγράψαμε πολλές φορές και προσθέσαμε και δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ε, το οποίο όταν υπάρχει ανάπτυξη σημαίνει μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην ε, ε, ωφέλει από αυτήν την ανάπτυξη και δεύτερον αυτό το μοντέλο πρέπει να ε, μεταφράζεται σε 26 διαφορετικά συστήματα. Εγώ είμαι Βέλγος, γνωρίζω πολύ καλά το βελγικό σύστημα, είναι διαφορετικό ακόμη και σε πολύ σημαντικά ζητήματα από τι οι γείτονές μας, οι πολύ κοντινοί γείτονές μας. Λοιπόν, ε, αυτό βεβαίως ε, θα εμπνεύσει και κάποιες από τις απαντήσεις μας. Και το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω και ενδεχομένως ε, να είναι αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος Ντράγκη. Βεβαίως πρέπει να θεωρήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο επί σημείων γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το προσδόκιμο ζωής έχει εξελιχθεί. Οι ανάγκες των οικογενειών έχουν εξελιχθεί. Η διακοινωνία έχει εξελιχθεί. Άρα υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης κάποιων στοιχείων του μοντέλου προκειμένου το σύστημα το οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε να είναι βιώσιμο. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Ξέρω ότι ήσασταν πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων εδώ στο Κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία. Ε, μιλάω λοιπόν σε έναν ειδικό, σε έναν εμπειρογνώμονα. Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε ανάπτυξη ε, και οι οικονομίες ε, εξελίσσονται. Είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε μία ε, συνεδρίαση στη Γενέβη με τον Πασκάλ Λαμή την περασμένη Παρασκευή, ο οποίος ειδικότερα σε σχέση με την Ευρώπη ανέφερε τον κίνδυνο για την έλλειψη ανάπτυξης σε, μία, σε ένα παγκοσμιούμενο περιβάλλον και συγκρίνοντας σε εμπορικό επίπεδο την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο ε, η απασχόληση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Πριν από την κρίση, ε, ναι, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, ε, οι επιχείρησεις όταν έχουν δυνατότητα εξελίσσονται αναπτύσσονται και εξορισμού, να δούμε τώρα βέβαια σε τι αναλογία το κάνουν αυτό, δημιουργούν άμεση και έμεση απασχόληση. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε σήμερα αν θέλουμε και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό, αν θέλουμε να έχουμε πιο υγιή δημόσια οικονομικά, θα πρέπει να αυξήσουμε τα ε, εισοδήματα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσω της ε, ε, φορολογίας, αλλά αν το κάνουμε μόνο με τη φορολογία, ούτε αυτό θα είναι βιώσιμο. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ειδικότερα στις χώρες όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμη πιο επισφαλής. Να δούμε την κατάσταση στη Γερμανία. Ξέρω πάντοτε έχουμε την Γερμανία ε, ως αναφορά. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία, τι να κάνουμε. Και είναι μια οικονομία που έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Παρά λοιπόν ε, την κρίση αυξάνεται η απασχόληση και μειώνεται η ανεργία παρά το γεγονός ότι είναι η χώρα η οποία μεταξύ των μεγάλων χωρών έχει τέλος πάντων το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης. Ε, νομίζω ότι υπάρχει κάποια σχέση, θέλω να πω υπάρχει πραγματική οικονομία για την οποία ομιλείτε. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση γιατί πάντοτε εμεί είχαμε υπερασπιστεί ε, το όφελο τη ανάπτυξη πραγματική οικονομία και στην πραγματική οικονομία, κυρία Πρόεδρε, συμπεριλαμβάνω και τον χρηματοπιστωτικό τομέα γιατί είδαμε ότι σε αυτόν τον τομέα, ε, ε, χωρί αυτόν τον τομέα δεν λειτουργεί η οικονομία. Είμαστε κατά τη κερδοσκοπία μεν, είμαστε κατά του του γεγονότος ε, ότι ε, πρέπει να υπάρχουν, ότι είμαστε κατά των καταχρήσεων στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όλα αυτά ναι πρέπει να τα ξαναδούμε. Για τον κύριο Κρίστενσεν. Σε ό,τι αφορά το πακέτο ανάπτυξης και πώς αυτό συνδέεται με την ουσιαστική συζήτηση, τη βασική συζήτηση που είχαμε με τα συνδικάτα, και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά φαντάζομαι ότι τον ίδιο συζήτηση είχατε και εσείς εδώ για τις πολιτικές ε, λιτότητας και πώς ε, συνδυάζονται με την ανάπτυξη. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δεν ε, μπορούμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ξέρετε και εγώ ως Βέλγος μιλώ ε, με τα λόγω γνώσεως, ξέρω τι κάναμε, τι αναγκαστήκαμε να κάνουμε στις δεκαετίες του 80 και του 90. Ταυτόχρονα όμως, πέρα από την λιτότητα, χρειάζεται ανάπτυξη και μάλιστα χρειάζεται έξυπνη ανάπτυξη. Κάποια κράτη-μέλη βεβαίως έχουν πολύ μικρότερα περιθώρια λεγμών από ότι άλλα. Ε, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και για να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις, ναι πρέπει να δημιουργήσουμε τις ε, κατάλληλες συνθήκε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο έδαφος για ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Και υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι, ανέφερα πριν ε, το ψηφιακό τομέα, αλλά είναι και ο ενεργειακός τομέας, όπου εκεί δεν χρειάζεται δημόσιες επενδύσεις, χρειάζονται όμως απεγνωσμένα επενδύσεις. Το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο όμως πρέπει να υπάρχει, να είναι ε, ορθά δοσμένο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές. Ε, επίσης θέλω να πω ότι οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη δεν θα δημιουργηθούν μόνο αν αυξάνοντας τους φόρους. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια στην εργασία, το flex security, ναι, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο. Είπατε, δεν υπάρχει ακόμη αυτή η ισορροπία. Ναι, να το ζητήσουμε Από ποιο πρίσμα το βλέπετε, ότι δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. σε όλους τους τομείς, της κοινωνικής προστασίας. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να κρατήσουμε την κοινωνική προστασία, όμως πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε κάποια στεξιωτικά συστήματα, να ξαναδούμε, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις Εργασία. και όσο φορά τις κατηγορίες των ε, συμβάσεων εργασία, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε διαφορετικές μορφές συμβάσεων εργασία. Πρόσφατα είχαμε και ε, μία σχετική εξέλιξη, ένα γεγονός ότι αφορά τους ε, προσωρινά απασχολούμενους ε, ή μάλλον για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Θέλουμε όμως πρώτα απ' όλα να δώσουμε έμφαση και να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες για την προσχώρηση στην αγορά εργασία. Δεν έχω αυτή τη στιγμή αριθμητικά στοιχεία να σας δώσω, αλλά πάνω από το ίμιση αυτών που αρχίζουν να εργάζονται με μια ειδική ε, σύμβαση μέσω γραφείων έδρας εργασίας τελικά καταλήγουν σε μια σταθερή ε, σύμβαση απασχόλησης. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος πρόσβασης στην εργασία. Η κυρία Κορνέλησαν επίσης μίλησε για το θέμα της φτώχειας μέσα στην εργασία και για τους αξιοπρεπείς μισθούς. Ναι, από την οπτική γωνία των εργοδοτών μπορώ να μιλήσω γενικά για τους εργοδότες, υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσει. Και βεβαίω δεν υποστηρίζουμε τέτοια φαινόμενα. Εμείς πάντως εν γέννη φρονούμε ότι η εργασία θα πρέπει να παρέχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Βεβαίω η έννοια του αξιοπρεπού εισοδήματο είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν κατώτατοι μισθοί. Θεωρούμε ότι η κατώτατη αυτή μισθή σε σχέση με ε, την εργασία που θα πρέπει να ε, επιτελέσει κανείς, αυτός ο κάτω μισθός πάντως δίνει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Η πάταξη όμως της φτώχειας που είναι από τους στόχους στρατηγικής του 2020. Εμείς τι είπαμε. Για να δούμε πώς θα επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ο καλύτερος τρόπος και πάλι είναι να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν μια θέση εργασίας. Εμείς ποτέ επί της αρχής δεν θα υπερασπιζόμασταν την ε, εργασία που παρόλα αυτά κρατάει τον άνθρωπο στη φτώχεια. Και τέτοιου είδου φαινόμενα δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ε, πολλοί εργαζόμενοι που από αυτούς εξαρτώνται παιδιά. Ε, και άρα είναι ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο που πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά τώρα. Για την αναντιστοιχεία των δεξιοτήτων, κυρία Κορνέλισεν, υπάρχουν στοιχεία εκπαίδευσης και για να απαντήσω και σε κάποιες άλλες παρεμβάσεις και ευχαριστώ όλους σας για αυτές, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να δούμε για να συνδέσουμε τους οικονομικούς πέκτες και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η, κοινό, η Κομισιόν πριν από χρόνια είχε αναλάβει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία σε ένα φόρουμ που είχε τίτλο «Πώς να φέρουμε κοντά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για να συνεργάζονται στενότερα οι δύο αυτό πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης και στην βάθμια εκπαίδευση. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό στοιχείο. Για τους μισθούς υπογραμμίζω και εγώ ότι στη Γερμανία θα αυξηθούν κατά 4% κατά μέσον όρο κατόπιν συμφωνιών οι μισθοί. Αυτό σίγουρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί πάντοτε στη Γερμανία αποφασίζονται με βάση συλλογικές ε, συμβάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα γίνει δεκτή συμφωνία, γιατί στηρίζεται στον κοινωνικό διάλογο. Κύριε Ορί. το να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσει απασχόληση. αυτό είναι το προφανές και το τονίζουμε και στις ε, θέσει ε, που λάβαμε ε, προσφάτως μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων. Έφτασε επιτέλους ο καιρό να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για ιδιωτικέ επενδύσεις. Ό,τι μπορούμε να ενθαρρύνουμε, όπως μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να το κάνουν, πρέπει να τι ενθαρρύνουμε. Θέλουμε όχι μόνο με φορολογικό τρόπο να το κάνουμε αυτό, κυρίως όχι με αυτόν τον τρόπο. Ε, να δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει η ιδιωτική σφαίρα. Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνουμε ε, κυρίως για τα επαγγέλματα υγείας, ε, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση του άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη, αλλά χωρί να τιμωρήσουμε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τις ε, μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην κυρία Γιασλοβίσκα, καλά τα πήγατε με την προφορά. Γιασλοβίτσκα. Ε, μίλησα για τους μισθούς. Ο, ως επιτοπλίστων είπα ότι πρέπει να μειώσουμε το κόστος εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να μειώσουμε τους μισθούς. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες, ε, λόγω των μνημονίων, πρέπει να γίνει μια ε, μείωση. Εκεί μιλάμε για λιτότητα. Αλλά η μείωση του κόστου και των εισφορών των εργοδοτικών, ε, αυτό νομίζω ότι είναι μια επένδυση. Τώρα, για τα, τις διάφορες μορφές συμβάσεων απάντησα και για την κατάρτιση, μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και ίσως θα πρέπει να γίνει δουλειά σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ε, πλησιάσει να πλησιάσουν μεταξύ του οι εκπαιδευτικοί και η επιχειρηματική κοινότητα, γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχει κάποια μεγάλη απόσταση και κενό ανάμεσά τους. Μιλήσατε για τα χρηματοδοτικά μέσα. Εμείς τα χρησιμοποιούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο γιατί είναι ε, επαχθείς και μεγάλες διαδικασίες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία γιατί αυτά τα μέσα είναι σημαντικά για μόχλευση και στο κοινωνικό επίπεδο. Συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ειδικής ε, εκπαίδευσης και της μαθητείας. Και για τα στάζ, που είναι και η τελευταία μου ερώτηση, νομίζω ότι ήταν και η τελευταία, η τελευταία μου απάντηση, γιατί είναι και η τελευταία ερώτηση, δεν νομίζω ότι τα στάζ μπορούν να θεωρηθούν ε, ω κοινωνικό dumping Οι κανόνες ε, αποφασίζονται, ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και για τα στάζ, αυτές τις περιόδους μαθητεία, ε, ε, όπως και σε άλλους κοινωνικούς τομείς, οι ελάχιστες προϋποθέσεις ε, δεν τις θέλουν ούτε τα συνδικάτα, γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι συνθήκες οι ελάχιστες που ζητάτε, οι προϋποθέσεις οι ελάχιστες που ζητάτε είναι τόσο διαφορετικός ε, σε διάφορες χώρες. Δεν θα έχουμε ποτέ τέτοιου είδους εντολή εμείς για να διαπραγματευτούμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτήν ε, λοιπόν ε, την διαπίστωση των ορίων ε, των κοινωνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι η τελευταία σας εμφάνιση στην, σημερινή, στην Επιτροπή μας, η σημερινή, μέχρι σήμερα και εδώ και με άλλες ευκαιρίες είχαμε πάντοτε επικοδομητικούς, ε, επικοδομητικές και ζωηρές ε, συζητήσεις ε, για αυτό το θέμα του οποίου είστε υπεύθυνο. αναπτύξατε αυτό που τότε ήταν πριν από την Business Europe η UNICEF Παραλίγο να το ξεχάσω. Πολύ καλό αυτό το, πολύ καλό σημάδι αυτό λέει ο κύριος The Book. Ναι, ε, πάρα πολύ συνεισφέρατε εσείς σε αυτήν την μετάβαση από τη UNICEF στην Business Europe. Ε, ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει τους διαλόγους μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ε, σε κάθε κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Καλή σας επιτυχία στην ε, συνέχεια των προσωπικών και ευρωπαϊκών σας περιπετειών και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που μας ε, συνόδευσαν μέχρι το τέλος των πρωινών μας εργαζιών γιατί θα ξαναρχίσουμε στις 3 η ώρα με την παρουσίαση της Κυπριακής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.